Buenos días a todos. Σας καλημερίζω όλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την συνεδρίαση της Επιτροπής μας με μια μικρή υστέρηση χρονική. Estoy coincidiendo con el café. Comenzamos con la aprobación. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει και μία σειρά θεμάτων που θα ήθελα να σας θέσω. Υπάρχει μία πρόταση αναβολής για την επόμενη συνεδρίασή μας των σημείων 4 και 5. Ψηφοφορία των σημείων 4 και 5. Ντόντους. Ένα τώρα. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχετε να θέσετε κάποιο άλλο θέμα, αλλά τα θέματα αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν στην επόμενη συνεδρίαση. Σχετικά με το 7 τώρα, για τη συμφωνία δηλαδή με τη Μαυριτανία. Από ορισμένε πολιτικές ομάδες έλαβα σαν εισηγητής την πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας μέχρι την επόμενή μας συνεδρίαση. Σας εξηγήσω γιατί. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση αναβολής είναι ότι ήδη υπήρξε μια συνάντηση της Μικτής Επιτροπής. Σε κάποια θέματα έχουν γίνει βήματα προόδου, σε άλλα λιγότερο. αλλά από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει σύγκληση μετά από αυτή τη συμφωνία της Επιστημονικής Επιτροπής. Η άποψή μου λοιπόν είναι σαφής. Εμείς θέλουμε μια συμφωνία με τη Μαυριτανία, Ξέρουμε ότι η συμφωνία αυτή ως έχει δεν έχει, δεν είναι ιδιαίτερα θετική και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουν να έχουν την θετική άποψη του Κοινοβουλίου εφόσον θέλουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ας υπάρξει λοιπόν κάποιος χρόνος για να υπάρξει μια κάποια συμφωνία και γι' αυτό προτείνω την αναβολή της ε, απόφασης μέχρι την επόμενη εβδομάδα με στόχο, όπως είπα, τη βελτίωση της συμφωνίας και την απόκτηση μια θετικής γνώμης από πλευράς του Κοινοβουλίου. Κύριε Στόρβαλτς συζητήσαμε το θέμα αυτό και θα μπορούσαμε να δεχθούμε την πρόταση ως έχει και το έχω ήδη πει αυτό. Στην περίπτωση ψηφοφορίας όμως σε αυτή τη φάση θα τηρήσουμε στάση αποχής κατανοώντας λίγο και τις απόψεις των υπολείπων πολιτικών ομάδων. Κατανοούμε λοιπόν την άποψή σα, αν και δεν τη συμμεριζόμεθα πλήρως, λέει ο κ. Στόρβαντ. Ευχαριστώ. Και εμείς θα θέλαμε να γίνει ψηφοφορία τώρα. Δεν νομίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιμένει για την ψηφοφορία αυτή γιατί κάτι τέτοιο πιέζει την Μαυριτανία μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής να ανοίξει ακόμα περισσότερο ε, <clears throat> τα δικαιώματα ενώ έχουν ε, υποσχεθεί στους αλληλείς τους για πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα. Ένα άλλο θέμα θέλω να θέσω κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό από ό,τι φαίνεται, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στην έκθεση για την Ευμαυριτανία, αλλά ούτε και στην έκθεση για τη Μαδαγασκάρη. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει άμεση διόρθωση. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Λάβινγκ σχετικά με την δυνατότητα ψηφοφορίας τώρα, ο κύριος Λογκαρέκ συγγνώμη. Ε, εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και θέλω να περιμένουμε την πρόταση της επιστημονικής... Η κυρία Ρόντος, προσωπικά θα ήθελα να πω, θα μπορούσα να ψηφίσουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια καινούρια πράγματα. Έχουμε μια απόφαση στην ομάδα εργασίας. Αν πρέπει κάτι να αναβληθεί, να αναβληθεί έστω. Γκαρθία Γέρο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω για αυτό το θέμα ο συνάδελφος Αντολίν έχει μια πιο αποκρισταλωμένη άποψη, αλλά δεν είναι παρόν. Θέλω να υποστηρίξω την άποψη και να συμμεριστώ την άποψη άλλων μελών της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής Όλοι εργαστήκαμε κατά τη διάρκεια πάνω από ένα μήνα τώρα και η δυνατότητα αυτή η Επιστημονική Επιτροπή να μπορούσε να εξετάσει τελικά μια λύση στο πρόβλημα το οποίο είχε τεθεί, μια και οι προϋποθέσεις που είχαμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά αυτό το ζήτημα είναι διαφορετική. Ζητήθηκε αναβολή σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται ούτε εδώ για το να πιεστεί ούτε η Βρετανία ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν υπάρχει όμως ε, εδώ η διαφορά όσον αφορά το θέμα της πίεσης για τα άλλα θέματα δεν είναι καθόλου πίεση. Είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο για να, έχουμε, να κάνουμε τα πράγματα με καλύτερο τρόπο. Αυτό πιστεύω πρέπει να κάνουμε σήμερα. Να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να αποφασίσουμε όχι υποπίεση αλλά για να γίνουν τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο. Να έχουν την καλύτερη έκβαση για όλους. Όχι μόνο για τα συμφέροντα ενός συμβαλωμένου, ή για, π.χ. για παράδειγμα για το Κοινοβούλιο, αλλά για όλους. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω και εγώ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρός μας, αλλά θα ήθελα να εκφράσω τις εξής σκέψεις. Μια συμφωνία πρέπει να είναι χρήσιμη για όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Τα χρήματα τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, θα έλεγα, ένα σημαντικό ποσό δεν έχουμε περάσει στη συζήτηση επί της ουσίας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις που κάνει. Και δεν είπε θα καταψηφίσουμε ούτε ο πρόεδρός μας. Δεν είπε να αναβάλουμε. Απλά έκανε μια πρόταση λογική λέγοντας ότι αν περιμένουμε την επόμενη συνάντηση της Επιτροπής θα πετύχουμε μια καλύτερη συμφωνία έτσι ώστε η συμφωνία αυτή να χρησιμεύει επαναλαμβάνω σε όλους. Να, ε, ε, εδώ επιστεύω την προσοχή των συναδέλφων σε αυτούς ε, που διαφωνούν ότι όχι ότι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε, αλλά θέλουμε να ψηφίσουμε καλύτερα και γι' αυτό χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες εβδομάδες. Ο κ. Μιλάνα Νομίζω ότι στην περίπτωση που ο εισηγητής ζητάει μια αναβολή για μια εβδομάδα θα πρέπει να το δεχθούμε καταρχήν. Είναι θέμα σεβασμού της προσπάθειας που κάνει ο εισηγητής. Αυτό ισχύει γενικά. Τώρα όταν αυτή η Επιστημονική Επιτροπή μπορέσει να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, <clears throat> δεν είμαι πολύ αισιόδοξο βέβαια, και εδώ θα υποφεληθώ της παρουσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας πει η Επιτροπή Εάν πράγματι πιστεύει ότι αυτή η συνάντηση στην οποία εμείς αποδίδουμε μάλλον μεγάλη σημασία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πει ότι κάτι τέτοιο θα είναι χρήσιμο, τότε αυτό είναι προς όφελος όλων και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Αν η Επιτροπή μας πει ότι η συνάντηση αυτή είναι άχρηστη σε σχέση με το θέμα το οποίο συζητάμε, ε, καλύτερα να ψηφίσουμε σήμερα. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε. Νομίζω θα συμφωνήσει ο Πρόεδρος μαζί μου. Λοιπόν, εφόσον αυτή η συνάντηση στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα κάτι δώσει, τότε να περιμένουμε, αλλιώ όχι. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή θέλει να μα δώσει κάποια ένδειξη, θα ευχαριστούσα. <clears throat> intervention Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Μια τεχνική επεξήγηση σε όλους. Αυτή η μεικτή επιστημονική επιτροπή πρώτον είχε σχεδιαστεί να διεξαχθεί σύμφωνα με την Μαυριτανία πριν από την κοινή επιτροπή της συνεδρίασης της στο Παρίσι. Αυτό δεν ήταν δυνατό επειδή δεν υπήρχε διαθεσιμότητα επιστημόνων των δύο μερών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε σε σχέση με τη Μικτή Επιτροπή για το Παρίσι. Κάνουμε λόγο τώρα για τη Μικτή Επιστημονική Επιτροπή για να μην υπάρξει κάποια σύγχυση. Τώρα, οι ημερομηνίε για τη Μικτή αυτή επιστημονική επιτροπή είναι από τη Δευτέρα έως την 5η Απριλίου. 2-5 Απριλίου, δηλαδή ε, σε δύο εβδομάδες. Ουσιαστικά από τεχνικής πλευράς η Μικτή Επιστημονική Επιτροπή είναι το σώμα εκείνο το οποίο εξετάζει οποιαδήποτε επιστημονικά θέματα σε οποιαδήποτε τέτοια θέματα ζωνών Συναπαρτίζεται και από τα δύο μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρατηρητής. Θα έχουμε τον επιστήμονά μας ή τους επιστήμονές μας ως παρατηρητές σε αυτή την μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή και η συμφωνία και των δύο μερών ανοίγει σε σχέση και με την συμμετοχή επαϊόντων εκ των έξω. Τώρα, τι μπορεί να κάνει αυτή η, μεικτή Επιστημονική ε, Επιτροπή. Να δει τα... τις διάφορες δυνατότητες αλληλείας, τα αποθέματα που έχουν σε σχέση με τα αλλιεύματα και να αξιολογήσει αυτούς τους όρους. Δεν θα ληφθεί κάποια απόφαση λοιπόν από αυτή την Επιστημονική Επιτροπή, διότι θα δώσει η Επιστημονική Επιτροπή μόνο συστάσεις τις οποίες θα συντάξει. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα υπάρξει μια νέα απόφαση που θα ληφθεί αυτόματα. Εντάξει, κάνω λόγο για οποιαδήποτε κατηγορία αλλιευμάτων και αλλιείας. Αυτό είναι σημαντικό διότι θα επικαιροποιήσει το πώς έχουν τα πράγματα από βιολογικής πλευράς. Αλλά να είμαστε σαφείς, αυτά όλα δεν θα καθορίσουν κάποιες τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις αυτόματα διότι είναι ένα επιστημονικό σώμα και το κύριο σώμα που σύμφωνα πάντα και μεταξύ ΕΕ και Μαυριτανίας μπορεί να λάβει κάποιες πιθανόν αποφάσεις είναι η Μικτή επιτροπή που ήδη διεξήχθη στο Παρίσι. Αυτή είναι η τεχνική επεξήγηση του τι θα συμβεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μέσνερ, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν δεν είχα ζητήσει τον λόγο διότι έχουμε τον σκιώδη εισηγητή μας στην Επιτροπή Αλίας. Είχα κάνει εγώ αυτή τη γνωμοδότηση και είμαι αναπληρώτρια ως μέλος. Φυσικά πίσω από αυτή τη γνωμοδότηση που συνέταξα και γνωρίζω ότι όπως προτείνεται τώρα εδώ για τη Συμφωνία Αλίας ε, θα σημαίνει κάποια αλλαγή. Μια αλλαγή για πιο αηφόρο τρόπο αλίας, αλλά και μια αλλαγή προς μια περισσότερο αναπτυξιακή πορεία που ακολουθούμε στην Ευρωβουλή γι' αυτό. Και αυτό είναι μια αλλαγή. Και θα έλεγα ότι για την αλία συνεπάγονται αυτά μια αλλαγή και πρόκειται για μια σωστή συμφωνία. Εγώ θα ήμουν υπέρ μια ψηφοφορία σήμερα. Αλλά όπω αναφέρθηκε και από συνάδελφο, συζητήθηκε το θέμα στην Άλτε και δείχνω κατανόηση αν θέλουν να έχουν μια εβδομάδα χρόνο. Φυσικά θα ήταν καλύτερο να μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε, αλλά με βάση την εναλλακτική αυτή λύση και αυτό μπορεί να προχωρήσει. Ευχαριστώ κύριο Ρομέρο, παρακαλώ. Ε, Σα ευχαριστώ για το θέμα που το δικαίωμα λήψης απόφασης για τα πλεονάσματα τα αλλιευτικά στη Μαυριτανία εξαρτάται ακριβώς από την Επιστημονική Επιτροπή της Μαυριτανίας και όχι της κοινή Επιτροπής ή της Επιστημονικής Νικτής Επιτροπής. Ως προς όλα αυτά θα έπρεπε να είμαστε λοιπόν πρόθυμοι για να γίνει αυτή η ψηφοφορία. Συγγνώμη που το ξέχασα. Αυτό έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, Πρόεδρε, με αυτό. Λοιπόν, είμαστε πρόθυμοι να προβούμε σε ψήφιση. Όμως, συμφωνούμε και με το έτοιμά σα για, αναβολή. Σάντσε Πρεσέντο, παρακαλώ, τελευταίο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι αυτή η συμφωνία επηρεάζει εννέα κατηγορίες αλλιευμάτων έγινε μια συνεδρίαση στις 18 και 19 Φεβρουαρίου όπου σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή όσον αφορά ε, αυτά τα αλλιεύματα έγινε μια αποστολή επιστολών και κρεμεί τώρα το θέμα σε σχέση με απάντηση. Υπάρχει και κάποια άλλη κατηγορία για τα κεφαλόποδα και εκρεμεί μια αξιολόγηση των αποθεμάτων. Από τις εννέα κατηγορίες λοιπόν έχουμε τέσσερις, στις οποίες αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πώς θα επιληθούν τα προβλήματα που τίθενται. Και αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά ότι αφορά την αξιολόγηση σε σχέση με το σύνολο της συμφωνίας. Καθώς πιστεύω ότι βρισκόμαστε ακόμα σε έγκαιρη χρονική στιγμή, θα προτιμούσα να αναμείνουμε το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Δευτέρας έως 5ης απριλιου και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την επίλυση αυτών των θεμάτων. Εν τέλει με αυτά τα θέματα δηλαδή. Πρόκειται για τεχνικά και οικονομικά θέματα και χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία ως πληροφορία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να δούμε αν προχώρησε η επίλυση των προβλημάτων που είχαμε. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο Πρόεδρε, για να έχουμε αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chair. I just wanted to ask you as a rapporteur if you are going... Λοιπόν, εάν πρόκειται να αλλάξετε τη θέση σας και να υπερψηφίσετε τις τροπολογίες μας, αυτό πρόκειται να γίνει εάν η Μικτή ε, Επιστημονική Επιτροπή μας δείξει ότι μπορούν να τροποποιηθεί η θέση της σε σχέση με το χταπόδι στη Μαυριτανία. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ρωτήσω για το πώς ε, θα τοποθετηθείτε, αλλά δύο προσαφηνήσεις για την ε, αναβολή αυτής της ψήφισης. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις για κανέναν. Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά ούτως ή άλλως και γι' αυτό δεν καθυστερούμε κανέναν και τίποτα. Έτσι λοιπόν όποιος θέλει να αλλιεύσει μπορεί να αλλιεύσει. Όποιος δεν θέλει δεν θα πάει να αλλιεύσει. Και η θέση μας αυτή τη στιγμή είτε λυθεί σήμερα είτε την επόμενη εβδομάδα στην επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής δεν έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις. Όμως πρόκειται για το εξή. αν ψηφίσουμε σήμερα και καταψηφίσουμε τη συμφωνία που είναι πιθανό να μπορεί να γίνει, δεν θα έχουμε πια συμφωνία και θα πρέπει να ξαναεξεταστεί. Αν αναβάλουμε δεν αλλάζει τίποτα. Υπό τους ίδιους όρους ε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, μια και εφαρμόζεται προσωρινά, δεν αλλάζει κάτι. Κερδίζουμε πολύ περισσότερο περιμένοντας τα αποτελέσματα παρά εγκρίνοντας αυτή τη στιγμή τώρα. Διαρωτώ με, τι είναι σε σχέση με την παράταση αυτή το νόημα. Η θέση μου ήταν ως εισηγητού να υπάρχει μια συμφωνία με τη Μαυριτανία και αυτή εξακολουθεί να είναι η θέση μου και αναφερόμενος προς την Επιτροπή, αυτή η Επιστημονική Επιτροπή δεν θα αποφασίσει πολιτικά κάποια αλλαγή ή οποιαδήποτε αλλαγή. Όχι, αλλά μπορεί να επηρεάσει το πώς θα ψηφίσουν πολλά από τα μέλη της Επιτροπής μας. Αν υπάρχει πρόοδος σε κάποια θέματα, ίσως ε, μπορεί αυτό να αλλάξει κάποια πράγματα. Όμως, μόνο όταν θα υπάρχει μια σαφής πρόοδος ε, στα θέματα που έχουμε εμείς ε, και θέλουμε να προχωρήσουν για τους αλληλείς εκεί επί τόπου. τώρα, να ψηφίσουμε ή να μην ψηφίσουμε. Νομίζω συζητήσαμε επαρκώς και η τοποθέτηση είναι σαφής. Η δική μου πρόταση πρόταση ως εισηγητού είναι να αναβάλουμε, να αναβάλουμε σε σχέση με το θέμα αυτό την ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε τι συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία όταν θα έχει διεξαχθεί η συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής από τις 2-5 Απριλίου. Συμφωνείτε? Λοιπόν, αυτό θα ψηφίσουμε τώρα, την αναβολή. Αναβολή της ψήφισης για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Υπέρ. Bien, en contra. Κατά. Abstenciones. Ποιες. Τρεις. Λοιπόν, εγκρίνεται η αναβολή τη ψήφισης για την επόμενη συνεδρίασή μα. 15 νομίζω υπέρ, 4 εναντίον, 3 αποχές. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 και εδώ έχουμε πάλι μια πρόταση αναβολής της ψήφισης ε, αυτού του σημείου για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Κύριε Ριβελίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες βέβαια, γιατί το θέμα που αφορά την εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μαδαγασκάρη στην Αλία επί της ουσίας θα έλεγα <clears throat> συναντά τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών ομάδων. Ο φάκελος λοιπόν ως έχει προτείνεται από όλους. Υπάρχει όμως συγκεκριμένα το αίτημα ιδιαίτερα από πλευρά της σοσιαλιστικής ομάδας και της ομάδας των Πρασίνων να αναβληθεί η ψηφοφορία για μετά τις εκλογές που θα γίνουν στη Μαδαγασκάρη. Λαμβάνοντας υπόψη Στη συνεργασία την οποία είχαμε ανάμεσά μας όλες οι πολιτικές ομάδες, θεωρώ ότι η πρότασή τους στα πλαίσια μιας τέτοιας συνεργατικής εισαγωγικά έκθεσης πρέπει να γίνει δεκτή. Είναι σαφές όμως ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο σημεία σήμερα πριν προχωρήσουμε ε, στην ε, συγκεκριμένη ψηφοφορία. Το πρώτο σημείο είναι ότι επί της ουσίας το θέμα αυτό μας βρίσκει όλους συμφώνους. Δηλαδή, ακόμα και αν εμείς αναβάλουμε για μετά από τις εθνικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη την εξέταση του θέματος, δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Γιατί επαναλαμβάνω ότι όλοι συμφωνούμε. Η πρόταση γίνεται λόγω ακριβώς των εκλογών, η πρόταση αναβολής. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι κατά. Ως εκ τούτου λοιπόν είμαι διατεθειμένος να αποδεχθώ την πρόταση των πρασίνων όπως και των σοσιαλιστών αλλά μέσως μετά τις εκλογές και αν δεν υπάρξουν ε, εξελίξεις αρνητικές στη Μαδαγασκάρη το θέμα θα πρέπει να γίνει δεκτό, η πρόταση θα πρέπει να γίνει δεκτή ομόφωνα όπως ε, ισχύει σήμερα. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση. Εμείς δεν αναλύουμε το συγκεκριμένο θέμα, το αναβάλουμε όμως και το ε, βάζουμε, αν θέλετε, να υπόκειται ε, στις πολιτικές, στις βουλευτικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη. Λοιπόν, έπρεπε να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα Επαναλαμβάνω ότι επί της ουσίας υπάρχει πλήρη συμφωνία και δέχομαι την πρόταση των σοσιαλιστών και των πρασίνων για μετά τις εκλογές στη Μαδαγασκάρη, αλλά με τις δύο διευκρινήσεις τις οποίες ήδη διευκρίνησα σε εισαγωγικά. Σύμφωνοι αποσαφινίστηκε. Η απόφαση είναι για την αναβολή στην επόμενη κοινοβουλευτική μας συνεδρίαση, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Εντάξει, για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έτσι, δεν ήταν απόλυτα σαφές. Τι συμβαίνει ακριβώς, με ποιες, εκλο... για ποιες εκλογές γίνεται λόγος. Αλλά μετά από τις εκλογές ή στην επόμενη συνεδρίασή μας. Τι λέτε κύριε Ριβελίνη. No, Για μετά τις εκλογές κύριε Πρόεδρε εγώ διευκρίνησα τις δύο αυτές λεπτομέρειες για μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη. Είμαστε σύμφωνοι λοιπόν, είναι σαφές. Ε, το αφήνουμε λοιπόν μέχρι μετά τις εκλογές όπως αναφέρθηκε. Και τέλος, όχι τέλος, υπήρχε κάτι άλλο. Όχι, είναι το τελευταίο, το σημείο 9 στην ημερησία διάταξη λοιπόν. Το 9 είναι η έκθεση του κυρίου Αρσένη. Σε αυτό το θέμα εγώ θέτω την τροποποίηση γι' αυτό δεν συμφωνούσε ο κύριος ε, Αρσένης, αλλά ίσως θα πρέπει να το δούμε αυτό. Η τοποθέτηση για την έκθεση αυτή είναι η τροποποίηση της ημερησίας διάταξης, όχι για να ενταχθεί σε άλλη συνεδρίαση, αλλά για να ενταχθεί στη συζήτηση αύριο, στο σημείο αμέσως μετά τη συνάντηση των συντονιστών μας αύριο. Για ποιο λόγο, για ένα απλό λόγο. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά λόγων, αλλά για ένα απλό λόγο. Πρώτα, πρώτα απ' όλα θα δούμε για, και την καθυστέρηση πάνω από ε, τον εύλογο χρόνο αυτή τη ε, μετάφραση δόθηκε στι 6 παρα 20 περίπου ε, ε χθε το βράδυ. Δεν είναι όμω ο μόνο λόγο. Ε, θα μπορούσε να ήταν και διαθέσιμη η έκθεση και πιο πριν σε κάποιες γλώσσες. Αλλά επειδή δεν ήταν όλες διαθέσιμες οι γλώσσες, γι' αυτό δεν διανεμήθηκε. Και τώρα λοιπόν πρέπει να ε, δούμε αυτό ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχει παράπονο λοιπόν, να μην υπάρχουν παράπονα για κάποιου που δεν θα είχαν τη μετάφραση στη γλώσσα του και άλλου που θα την είχαν. Αυτό είναι ένα λόγο, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ε, πήρα μια επιστολή από πλευρά 10 ε, βουλευτών που κάνουν μια παρέμβαση για την πιθανή ακρόαση για τις επιχειρήσεις ή αλληλείς ή και κάποιο βουλευτή την κυρία Τόμας ε, σε σχέση με ε, συναφή θέματα. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν στη συνάντηση των συντονιστών όμως. Νομίζω ότι είναι πιο λογικό η συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Αρσένη να γίνει μετά τη συνάντηση των συντονιστών λοιπόν όταν θα έχουν υιοθετήσει τις αποφάσεις που πρέπει να αποφασίσουν αύριο και έτσι να συζητήσουμε μετά την έκθεση του κυρίου Αρσένη μετά το να το κάναμε πιο πριν, πρώτον θα μετέτρεπε τη συζήτηση για αυτή την έκθεση σε άλλη σειρά θεμάτων τελείως διαφορετική ε, από πλευράς φύσης ε, ε, σε σχέση με τα θέματα και για την λήψη απόφαση πάλι θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα στη συνέχεια μετά τη συνάντηση των συντονιστών. Είναι πολύ πιο λογικό να ακούσουμε πρώτα του συντονιστέ τι αποφασίζουν και μετά να εξετάσουμε και να συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Αρσένη. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει στην ίδια συνάντηση αυτή τη επίτροπή. Δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση για τη διαβίβαση του φακέλου ή της έκθεσης αυτής. Και νομίζω είναι καλύτερο για όλους. Αυτή είναι η τη εκθεση αυτη και νομιζω ειναι καλυτερο για ολου αυτη ειναι η λογη για του οποίου ζητώ την τροποποίηση αυτού του σημείου στην ημερήσια διάταξη. Και από το 9 περνάμε στο 17 νομίζω. Μετά ακριβώς από συνάντηση των συντονιστών. 17α ή 17β θα γίνει. Ο κύριος Αρσένης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, με εκπλήσει λίγο αυτή η απόφαση γιατί η έκθεση μου είναι διαθέσιμη. Η έκθεση που έχει δοθεί, ε, έχει υποβληθεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να αναβληθεί η ψηφοφορία και όπως είπατε κι εσείς αντιτίθεμαι σφόδρα. Οτιδήποτε θα μπορούσε να συζητηθεί με τους συντονιστές, δεν πρόκειται να αλλάξει το περιεχόμενο της έκθεσης η οποία έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και στο κοινό. Επομένως, αντιτίθεμαι στην πρότασή σας. Ευχαριστώ. Λοβίν, παρακαλώ, η κυρία Λοβίν. Θυμάμαι, νομίζω ότι είναι στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής που ο πρόεδρος είχε πει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση να αλλάζουμε συνέχεια την ημερήσια διάταξη και είχατε πει ότι θα ε, πάψετε να το κάνετε αυτό παρά μόνο αν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Για λόγους διαφάνειας, μιας και επιθυμούμε η Επιτροπή μας να λειτουργεί με διαφάνεια, θέλουμε ο κόσμο να μπορεί να κοιτάει την ημερήσια μα διάταξη στο ίντερνετ, να παρακολουθεί τη συνεδρίαση μέσω του web stream. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη δεν δίνει καλή εικόνα. Ο εισηγητής έχει προετοιμάσει την παρουσίασή του, έχει υποβάλει την έκθεσή του. Οι ε, σκιώδες εισηγητές είναι επίσης παρόντες και θα ε, μπορούσαν να παρεύουν. Επομένως δεν βλέπω τον λόγο να μην συζητήσουμε την έκθεση ως έχει αυτή τη στιγμή. Και μετά στη συνάντηση των συντονιστών να συζητήσουμε οτιδήποτε ε, απομένει. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, άκουσα την θέση της κυρίας Λοβέν. Και θυμάμαι αυτό που είχατε πει για την ε, σημερινή στις αλλά οι πράσινοι θεωρούν ότι στο συγκεκριμένο θέμα γνωρίζω ποια είναι η θέση του κυρίου Αρσένη, οι συντονιστές δεν μπορούν να αλλάξουν την ουσία της έκθεσης, αλλά η έκθεση δεν είχε μεταφραστεί και δεν είχε διανεμηθεί, που μάλλον έχει διανεμηθεί. Εμείς όμως έχουμε και έχοντα υπογράψει την επιστολή που εστάλει στον Πρόεδρο, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιχειρήματα, ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά, για να δώσει στην ε, Επιτροπή, στα μέλη τη επιτροπή τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίε. Με την συνηθισμένη διαδικασία αυτή τη επιτροπή, πρέπει την απόφαση αυτή να τη λάβουν οι συντονιστέ και όχι η Επιτροπή στο σύνολό τη. Άρα μου φαίνεται λογικό να αναβάλουμε την απόφαση μέχρι αύριο. Δεν ζητάμε να αναβληθεί η συζήτηση για δύο και τρεις μήνες. Λέμε μόνο να αναβληθεί αυτό μέχρι να λάβουν οι συντονιστέ την απόφαση για μια πιθανή ε, επιπλέον ακρόαση. Έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε τι τροπολογίε έχοντα γνώση των γεγονότων πλήρη. Ευχαριστώ κύριος Μιλά. Εμένα η κατάσταση αυτή με εκπλήσει και σε επίπεδο αρχής ισχύει αυτό το οποίο ακούστηκε προηγουμένως. Η επιθυμία του εισηγητή σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι κυρίαρχη. Ακριβώς αυτό είπαμε και πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εισηγητή ζητήσει την αναβολή μιας ψηφοφορίας δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Αν πει ότι πρέπει να συζητηθεί σήμερα θα πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Πέραν αυτού όμως οι απόψεις τις οποίες εξέφρασε σαν παράδειγμα ο κύριος Στίβενσον μόλις προηγουμένως ε, είναι θα έλεγα κάτι το προφανές. Αν πράγματι συζητήσουμε σήμερα σαν παράδειγμα θα είχαμε τη δυνατότητα να ε, πάρουμε αποφάσεις ε, καλύτερα ενημερωμένοι, όχι. Νομίζω ότι θα είναι μία περίοδος χρόνου την οποία δεν θα εκμεταλλευτούμε, θα έλεγα, δεν θα, δεν θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Είναι επικίνδυνη η αναβολή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και δεν είναι δυνατόν μία, θα έλεγα, συνάντηση συντονιστών να τροποποιεί το πρόγραμμά μας με τον τρόπο αυτό. Είμαι κατά της προτάσεως αυτής λοιπόν επί της ουσίας. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση επί της ουσίας η συνάντηση, η συνεδρίαση των συντονιστών να τροποποιήσει και να αλλοιώσει την ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή, αν δεχθούμε την πρόταση, δημιουργούμε μία ιεράρχηση ανάμεσα στην συνάντηση, την συνεδρίαση των συντονιστών από τη μία και στην ολομέλεια της Επιτροπής μας από την άλλη. Η κυρία Ρόντοστ, ευχαριστώ πολύ και στην αρχή θα παρέμβω. Για να το ε- εκφράσω προσεκτικά, είμαι έκπληκτη. Είμαι έκπληκτη πρέπει να πω. Έχουμε μια διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο και λέει αυτή η διαδικασία ότι ο εισηγητής κατά κανόνα <clears throat> με τους συναδέλφους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων πρέπει να συζητήσει πώς θα διαμορφωθεί μια κρόαση. Και αν έχω πληροφορηθεί σωστά, όλοι, όλες οι ομάδες είπαν ότι συμφωνούν συμφωνούν. Αυτούς που θέλουμε να προσκαλέσουμε, που ζήσαμε στην ακρόαση να τους προσκαλέσουμε ή αυτούς που προτάθηκαν. Έχω μια υποψία τώρα. Στην ακρόαση για τον ένα ή άλλο συνάδελφο ίσως δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα σαν αυτό που ανέμεναν. Και τώρα γίνεται η προσπάθεια με μια δεύτερη ακρόαση να δώσουν μια νέα, να υπάρξει μια νέα άποψη που θα αποκρισταλωθεί. Διαφορετικά θα συνέβαιναν τα πράγματα αν ο εισηγητής χωρίς να το ανασυνδέσει αυτό την ακρόαση την διοργάνωνε ο ίδιος αλλά δεν το έκανε αυτό οι άλλες ομάδες ε, συμφωνούσαν τώρα ο εισηγητής συνέταξε μια έκθεση οι συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες και είναι δυνατόν, είναι δυνατόν η έκθεση σήμερα να παρουσιαστεί Όσο είμαι μέλος σε αυτή την Επιτροπή δεν το έζησα ποτέ όταν είχε συνταχθεί και ήταν έτοιμη μια έκθεση να αναβάλλεται και να μην ε, συζητείτε και να μην εγκρίνετε επειδή χρειάζεται λέει μια δεύτερη ακρόαση. Η Ζαμπέλα Λεβίν έχει δίκιο κατά τούτο. Η ημερήσια διάταξη είναι δημόσια, μπορούν να προσέλθουν κάποιοι φιλοξενούμενοι. Ίσως και εδώ σήμερα στη συνεδρίαση υπάρχουν κάποιοι που ήρθαν για να ακούσουν ειδικά τις απόψεις του εισηγητή για αυτό το θέμα. Εμείς τι θα πούμε δεν μας ταιριάζει θα πούμε, δεν μας γουστάρει, χρειαζόμαστε δεύτερη ακρόαση. Είμαι κάθετα εναντίον και θα το πω στη συνάντηση των συντονιστών. Νομίζω έχει κάθε δικαίωμα ο εισηγητής Αρσένης να παρουσιάσει σήμερα εδώ και τώρα την έκθεσή του. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Προτού συνεχίσω να δίνω τον λόγο σε μέλη, ένα θέμα. Επειδή ακριβώς συζητάμε αυτό το οποίο πρότεινα να μην συζητήσουμε. Και έτσι το δηλώνω αυτό, το λέω. Συζητείται εδώ η δυνατότητα να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Δεν συζητάμε άλλη ακρόαση ή όχι. Αν είναι πιο λογικό να κάνουμε το ένα ή άλλο, αν πίστηκε ο ένας ή ο άλλος ή τι πρέπει να γίνει. Δεν θα συζητήσουμε αυτά. Ούτε πρέπει να συζητηθούν σε σχέση και με την έκθεση. Αυτό προσπάθησα να αποφύγουμε. Εδώ σε καμιά στιγμή δεν τέθηκε το θέμα του ότι οι συντονιστέ λέει υποκαθιστούν ή θα πρέπει να αποφύγουν να υπάρξει μια συζήτηση. Με κανένα τρόπο. Το μόνο το οποίο ζητήθηκε είναι απλώς να πούμε για να μην δεσμευτεί κανείς με κανένα τρόπο η συζήτηση να γίνει μετά την λήψη απόφαση των συντονιστών. Γιατί, διότι μετατρέπεται η συζήτηση όπως μετατράπηκε τώρα σε μια συζήτηση γιατί έγινε το ένα, γιατί το άλλο και για την ουσία της πρότασης που επαναλαμβάνω είναι η έκθεση του κυρίου Αρσένη που προφανώς ε, ε, έχει κατατεθεί και όλοι την έχουμε αληθεύει ότι λίγο αργότερα θα πρέπει αυτά τα θέματα να μπορέσουν να προσαφινιστούν. Μια και έχουν ζητήσει και άλλοι τον λόγο, πρέπει να σας πω ότι δεν θα αφήσω σε αυτό το θέμα να γίνει λόγος για, το, για την ακρόαση, γιατί το ένα ή γιατί το άλλο. Απλά και μόνο θα συζητήσουμε τον, την τροποποίηση ή όχι τη ημερήσιας διάταξης, αναβάλλοντας σε ένα άλλο σημείο 17α την έκθεση του κυρίου Αρσένη, μετά τη συνάντηση των συντονιστών. Και, να, και θα δούμε σε ποιο σημείο θα είναι, στο, μετά το 17 ε, ε, ή όχι. Ε, αν παίξουμε καθαρά το παιχνίδι θα πρέπει όλοι να τηρήσουμε τους κανόνες και με κατανοεί απόλυτα ο κύριος Αρσένης. Άκουσα πριν λίγο ότι πάντα ζητούμε την άποψη του εισηγητή. Θα ήθελα πρώτα να υπενθυμίσω ότι η συζήτηση για το Ταμείο Αλίας έχει αναβληθεί πάρα πολλέ φορές χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή. Εκεί δεν ακολουθήσαμε την ίδια τακτική. Τώρα, η πρόταση του Προέδρου, ε, λυπάμαι, αλλά έτσι έχει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, θεωρώ ότι είναι προσβλητικό να ακολουθεί κανείς τέτοια επιχειρήματα. όταν ήμουν εισηγητή, αποφασίσατε να αναβληθεί η συζήτηση για την εκθεσή μου χωρί να υπάρχει σύμφωνη γνώμη μου. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα επιχειρήματα του Προέδρου είναι σωστά. Δεν ζητάει και τίποτα άλλο παρά να περιμένουμε μετά τη συνάντηση του συντονιστών αύριο και μετά θα γίνει μια σωστή συζήτηση και με τον κύριο Αρσένη. Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρία τέταρτα και έχουμε φτάσει στο σημείο εννέα υποτίθεται. Έχουμε αναβάλει τις αποφάσεις σε όλα τα προηγούμενα θέματα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής όχι για πάρα πολύ καιρό, αλλά παρόλα αυτά μένω σε παράκτιες περιοχές ε, με αλλιευτικές δραστηριότητες. Έρχομαι εδώ όπου λαμβάνονται αποφάσεις και τώρα έχω αρχίσει και καταλαβαίνω γιατί τα πράγματα πάνε στραβά. Και δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην επαναπατρίσουμε τα θέματα της αλλιευτικής πολιτικής στη χώρα μου. Αν δεν συζητάτε τίποτα πια. Κύριε Ντέιβις. Ευχαριστώ. Έχω κάποια πραγματικά εξαιρετικά επιχειρήματα, τα οποία όμως δεν θα, δεν θα πείσουν ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Ας τα θέσουμε σε ψηφοφορία παρακαλώ. Ο κύριος Αντινόρο. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους συναδέλφους. Να πω ότι είναι πρώτη φορά που πριν από την ψηφοφορία συζητάμε τόσο πολύ καιρό τόσο πολλή ώρα, 50 λεπτά. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ. Θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Γνωρίζω ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του συναδέλφου Μιλάνα. Κάποιοι από εμά είμαστε μέλη της Επιτροπής και συντονιστέ των πολιτικών μας ομάδων. Πριν έρθουμε λοιπόν εδώ, ε, ο καθένας συνεδριάζει με τα μέλη της ομάδας του, συλλέγει τις θέσεις, ε, ε, λιένει τις αντιπαραθέσεις και στην ουσία είναι θα έλεγα οι φωνές των πολιτικών του ομάδων, οι συντονιστές. Αυτό το, το λέγω για να θυμίσω και στον εαυτό μου το πώς δουλεύει το σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση του Προέδρου, η οποία είναι μια πρόταση η οποία έχει ανεπίσημα συζητηθεί και με άλλες πολιτικές ομάδες, έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι αύριο το πρωί στην συνάντηση των συντονιστών θα ξαναγίνει μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και από αυτήν την συζήτηση θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος της αποφάσεις και ε, θα ακολουθήσουμε ανάλογα. Ζητάμε μία αναβολή λοιπόν 24 ώρων και όχι 24 μηνών και είναι έλογο στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνουμε δεκτή την έκκληση του Προέδρου στα πλαίσια της λογικής και της βελτιωμένης λήψης απόφασης. Ευχαριστώ κύριε Τόμας. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais donc pas parler du... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς και δεν θα μπω στην ουσία, αλλά αλλά προσωπικά σας είχα ζητήσει εδώ και πολλές εβδομάδες, εάν ήταν δυνατόν, να γίνει μια μελέτη αντικτύπου κοινωνικο-οικονομικού, εάν αύριο οι συντονιστές αποφασίσουν κάτι τέτοιο, αυτό θα με ικανοποιήσει ιδιαίτερος. Δεν μιλώ για ακρόαση, αλλά έχουμε συζητήσει πολλές φορές ποιο είναι το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά δεν κοιτάμε ποιο είναι ο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Πολλοί, πολλά μέλη έχουν, είχα, έλαβαν το λόγο στην ακρόαση για να θέσουν αυτό το θέμα. Άρα, ελπίζω οι συντονιστέ να έχουν τη δυνατότητα να το συζητήσουν και να λάβουν σχετική απόφαση. Κύριε Ρομέβα, παρακαλώ. Ε, για να απαντήσω στον συνάδελφο την κυρία Καντέκ. Καμία σχέση. Ε, εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα τα οικονομικά ζητήματα. Ε, λοιπόν, ήταν σαφέ. Θα επικεντρωθούμε στην αλλαγή, όχι σε άλλη συζήτηση. Ο εισηγητή σήμερα είναι εδώ, όλοι έχουμε έρθει εδώ για να συζητήσουμε, έχουμε το κείμενο στα χέρια μας και δεν βλέπουμε γιατί να το αναβάλουμε τη συζήτηση. Γιατί, τι θα κερδίσουμε με το να αναβάλουμε τη συζήτηση αύριο. Ο εισηγητής είναι εδώ και είναι έτοιμος, δεν βλέπω γιατί. Ε, βοηθάει η αναβολή. Ο Ριβελίνη, eh, Πρόεδρε, αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη φάση είναι θα έλεγα κάτι το αρκετά σημαντικό και το οποίο έχει κρατήσει βέβαια πάρα πολύ ώρα όπως είπε ο Βρετανός συνάδελφος. Ε, θα έλεγα ότι εδώ και τέσσερα χρόνια δουλεύουμε πολύ σωστά και τώρα βλέπω να έχουμε μπλοκαριστεί. Ξέρω ότι αύριο καλό θα είναι να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και τους κανόνες λειτουργίας μας. Αν δεν έχουμε κάποιους γενικούς κανόνες λειτουργίας, θα ερχόμαστε κάθε πρωί εδώ και για 40-50 λεπτά θα συζητάμε για θέματα που δεν ενδιαφέρουν πράγματι καθόλου αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με μας. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τους κανόνες, θα πρέπει να σεβαστούμε την συμφωνία κυρίων που έχουμε Συμφωνώ με τον κύριο Λουκαντέκ, ε, δεν είμαστε εδώ ε, μία σκέτη πολιτική ομάδα. Θα ήθελα να πω στην κυρία Λεωδίν αυτό που λέμε εμείς στην Ιταλία, εξαιρετική συνάδελφος. Μην κάνεις ποτέ στους άλλους αυτό το οποίο ε, δεν θέλεις να σου κάνουν. Δηλαδή, ε, ή έχουμε κάποιους κανόνες και οι κανόνες αυτοί είναι γενικής χρήσεως και κάθε φορά δεν θα πρέπει να αλλάζουμε τους κανόνες για να βολέψουμε τη μία πολιτική ομάδα ή από την άλλη. Μιλάμε τώρα για μία αναβολή 24 ωρών και σε 24 ώρες δεν γίνονται επαναστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, άκουσα όλες τις απόψεις. Και θέλω να προσαφηνήσουμε ένα θέμα σε σχέση με την κυρία Λέβιν. Διότι αληθεύει, έχετε ε, δίκιο. Είμαι πάντα υπέρ του να μην υπάρχουν τέτοιε αλλαγέ. Αλλαγέ. Ε, δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα, θέλουμε να δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα και έχουμε τα θέματα των αλλαγών. Αλλαγών σε σχέση με ε, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Όχι επειδή κάποιο ε, ε, είτε καθυστέρησε είτε όχι, δεν είναι όμω αυτά τα θέματα τη συζήτηση. Αν υπάρχει αυτή η αλλαγή είναι για λόγου που τεκμηριώνονται και δικαιολογούνται επαρκώ, αλλιώ δεν θα είχε ζητηθεί. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Ριβελίνη, οι κανόνε δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι η πολιτική αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων που έχουν περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρον. Ή επειδή κάποιο μπορεί να νομίζει ότι σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να γίνει κάτι ή όχι. Σε σχέση με αυτό το θέμα, με κανένα τρόπο δεν ε, δεσμεύεται κάτι, δεν ε, τροποποιείται κάτι με την αλλαγή τη απόφαση σε σχέση με τη συνάντηση των συντονιστών. Θα έχει συνταχθεί η έκθεση, θα συζητηθεί το θέμα και θα δοθεί συνέχεια. Άλλο διαφορετικό θέμα είναι ο καθένας ε, να μπορεί να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα. Σε αυτή την Επιτροπή ε, είχαμε ε, σημαντικά θέματα διότι δύο μέρες, ε, τρεις μέρες όταν είχε κατατεθεί μια έκθεση μεταφρασμένη σε κάθε μια από τις γλώσσες και τώρα σε 14 ώρες ε, είναι κάτι το καταπληκτικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μια έκθεση 50 σελίδων ε, να είναι στη διάθεσή σας ε, μέσα σε 14 ώρες. Τώρα, δεν συμβαίνει το ίδιο σε σχέση με θέματα τα οποία εξυπηρετούν κάποιους κάποια, κάποια χρονική στιγμή να συνεχίσουμε τους ίδιους κανονισμούς. Ελάχιστες αλλαγές όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Χωρίς αμφιβολία. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτά γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κατά τη διάρκεια όλων των, ε, όλης της περίοδου προσπαθήσαμε να μην γίνονται τέτοιες αλλαγές. Ακριβώς επειδή το Συμβούλιο, η Επιτροπή, οι πολίτες ε, ε, ενημερώνονται για, την, για αλλαγές που πολλές φορές με πολύ λιγότερους λόγους τεκμηριώνονται από σήμερα αυτή η αλλαγή. Νομίζω επαρκώ έχει συζητηθεί το εξεταστεί το θέμα, επαναλαμβάνω. Έγινε λόγο για κάποια θέματα τα οποία αφορούν την ψηφοφορία ή για μια δεύτερη ακρόαση ή προθεσμία τροπολογιών. Δεν πρόκειται για αυτό. Θα γίνει η εξέταση θα γινει η εξεταση οπω σε σχέση με όλε τι εκθέσει και όλε τι συζητήσει. Απλά όμω, αντί για το σημείο 7 ή 8 που είχε προβλεφθεί η έκθεση, το 9, αντί το 9 συγγνώμη θα περάσουμε στο 17 μετά τη συνάντηση των συντονιστών. Και έτσι θα διατηρηθεί αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Διότι θέλουμε να τηρούμε τον λόγο όταν ε, έχουμε δεσμευτεί ε, και την υπόσχεσή μας. Περνάει λοιπόν το σημείο από το 9 στο 17 μετά τη συνάντηση των συντονιστών. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Καμία. Τροποποιείται λοιπόν η ημερησία διάταξη όπως είχε ζητηθεί. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα σε σχέση με την ημερησία διάταξη. Ευτυχώς κιόλα. Και περνάμε αν συμφωνείτε στην έγκριση τώρα των πρακτικών. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε τη μετάφραση των πρακτικών της 21ης και 22ης που δεν ήταν ε, διαθέσιμες για 18 και 19 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η έγκριση των πρακτικών μέχρι αυτή τη σημερινή συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις και του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, τα πρακτικά τους θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις ως ήθιστε μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας σήμερα. Από την άλλη πλευρά μας ε, στο σημείο 3, ανακοινώσεις του Προέδρου, συγγνώμη. Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας μας ενημέρωσε, συγγνώμη, συνεχίζει τις εργασίες της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Παρακαλώ ησυχία. Ξέρω ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν δίνουν σημασία. Αλλά παρακαλώ ησυχία, πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, η Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας ε, μας ανακοίνωσε ότι λόγω νέου ωραρίου της διάσκεψης των Προέδρων, νομίζω στις 3 το απόγευμα, λείπει η διερμηνία προς τα Δανέζικα. Δεν έχουμε διερμηνία προς τα Δανέζικα. Όμως έχουμε παθητική διερμηνία από τα Δανέζικα. Μπορείτε να μιλήσετε Δανέζικα και αν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να μιλήσει Δανέζικα και θα διερμηνευθεί. Επίσης ανακοινώνω ότι έχουμε την επίσκεψη μιας σημαντικής αντιπροσωπείας σήμερα από την Ισλανδία, χώρα που όσοι ήθιστε είναι παρούσα σε αυτή την Επιτροπή Αλίας και παρακολουθεί τις εργασίες. Και σε σχέση με την Αλία είναι πολύ σημαντική αυτή η συνιστόσα. Έχουμε αυτή την επίσκεψη με πέντε μέλη από την Ισλανδία. Ασμούντουρ, Όλαυσον, Όλριχ και Χιάλτα Δοδίρ. Συγγνώμη αν πρόφερα λάθο τα ονόματά σα. Καλώ ορίσατε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είμαστε υπερήφανοι που είσαστε ανάμεσά μα ε, κατά τη σημερινή μα συνεδρίαση. Χωρί να καθυστερήσουμε άλλο, περνάμε αμέσω στην ψήφιση. Al punto número... Περνάμε αμέσως λοιπόν στο σημείο 6 που είναι ακριβώ οι αλλιευτικέ δυνατότητε οικονομική αντιπαροχή σε σχέση με τη Συμφωνία Σύμπραξη Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία Μαυρικίου. Ψηφίζουμε λοιπόν το ψήφισμα ω έχει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Είναι πολύ εύκολο να σηκώνουμε τα χέρια. Μαυρίκιο ψηφίζουμε. Εντάξει το είπα. Ναι, κυρία Λόβιν, συγγνώμη, η κυρία Λόβιν. Συγγνώμη, εσείς κυρία Λόβιν. Ήθελα απλώ να πω ότι στην αγγλική διερμηνία είπαμε Μαυριτανία και όχι Μαυρίκιο. Μαυρίκιο, για το Μαυρίκιο ψηφίζουμε. Δεν ξέρω αν ήταν δικό μου σφάλμα. Εν πάση περιπτώσει, Μαυρίκιο είναι. Εντάξει, το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Λεβίν θέλει τόσο πολύ να <laughs> διευθετηθεί το θέμα τη Μαυριτανία. Ακούει Μαυριτανία. Είναι το 6 για το Μαυρίκιο όμω. Ψήφι υπέρ. Τα. Αποχές. Καμία αποχή εγκρίνεται λοιπόν. Πολύ καλά. No, dije que era como era una única votación. Eh, entonces, el ponente recomienda. Δίνει λοιπόν σύσταση να εγκριθεί η σύσταση του πρωτοκόλου. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το 10 που είναι η ψήφιση για τη στρατηγική σε σχέση με την αλληλεία. Όχι, λάθος έκανα, συγγνώμη. Una votación más, porque Madagascar se ha... Έχει αναβληθεί και το θέμα της Μαδαγασκάρης, οπότε δεν έχουμε άλλη ψήφιση. Δεν ψηφίζουμε τίποτα άλλο, ωραία. Ε? Δεν έχουμε καμιά άλλη ψηφοφορία. Ολοκληρώσαμε. Περνάμε στο σημείο 10 τώρα. Κανονικό σημείο 10. Στρατηγική για την αλληλεία στην Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. Εισηγητής είναι ο κύριος Μιλάνα διατηρήσαμε κατά το Δεκέμβριο, είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα δώσουμε τον λόγο άμεσα στον κύριο Μιλάνα για να μας ενημερώσει, να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί έχουμε πολύ χρόνο για να συζητήσουμε την έκθεσή μου. Οπότε μπορώ να μιλάω πολύ ώρα κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι. Συμφωνώ και για τον Βρετανό συνάδελφο. Για μια στιγμή λέει ο Πρόεδρος. γιατί ο συνάδελφος αυτός από τότε που είναι μέλος επιτροπής μας έρχεται, ακούει την ε, ημερήσια διάταξη και μετά φεύγει αφού μας κάνει και κάποια μαθήματα συμπεριφοράς, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που είπα θα βελτιώσει τη φιλική μου σχέση με το συγκεκριμένο κύριο στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, Είχα και εγώ, θα έλεγα, είχα σκεφτεί να ζητήσω την αναβολή της συζήτησης, αλλά τελικά αποφάσισα να μην το κάνω. Γιατί όπως είδα έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα τον μήνα Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας, όπως γνωρίζετε, η οποία αφορά, θα, έλεγε, θα έλεγα, μια πειραματική προσπάθεια να δούμε τις θάλασσές μας με διαφορετικό τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα. Quanto per cercare di capire se esiste la possibilità di costruire all'interno nostra το θέμα είναι να προσπαθήσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουμε την δυνατότητα, θα έλεγα, μιας μεγάλης περιοχής σωστά καθορισμένης, συγκεκριμένη περίπτωση της Ανδριατικής θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ ευρωπαϊκές χώρες, μη ευρωπαϊκές χώρες και χώρες οι οποίες είναι στην πορεία για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξει στα πλαίσια δηλαδή μια προοπτικής ευρύτερης για την περιοχή η εφαρμογή των κανόνων της αλληλείας όπως υπάρχουν σήμερα και να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για να πειραματιστούμε θα έλεγα σε μια σειρά επιπλέον κανόνων. Οι κανόνες αυτοί στην ουσία αναγνωρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των, αυτής της περιοχής. Πρώτον, πρόκειται ε, για μια κλειστή σχετικά θάλασσα είναι για μια περιοχή θαλάσσια η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μορφολογικά διαφορετικά από την υπόλοιπη Μεσόγειο και από τις υπόλοιπες μεγάλες ε, θάλασσες. Η συνύπαρξη, όπως είπα, κοινοτικών χωρών, μη κοινοτικών χωρών και χωρών ε, σε διαδικασία ένταξης δημιουργεί έναν χώρο, θα έλεγα, ιδιαίτερα κατάλληλο έτσι ώστε να πειραματιστούμε θα έλεγα και σε επίπεδο ε, διεθνών συμφωνιών ανάμεσα σε γειτονικές χώρες και περιοχές, να συζητήσουμε επίσης και θέματα τα οποία αφορούν γενικότερα την Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή όπως είπα όπου υπάρχει μια διαφορετική ιστορία και μια διαφορετική μορφολογία από ό,τι στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν οι ρυθμίσεις ειδικέ για τη Μεσόγειο πώς εφαρμόζονται εκεί. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να ορίσουμε ένα χώρο και στα πλαίσια του χώρου αυτού να προγραμματίσουμε μια σε εισαγωγικά χωροτακτική προσπάθεια ορισμού των θαλασσίων περιοχών και να προσπαθήσουμε ακόμα και σε νομοθετικό επίπεδο να καταστήσουμε συμβατές τις προσδοκίες των αλλιέων, να διασφαλίσουμε την διάρκεια της συγκεκριμένης αυτής δραστηριότητας και την ικανότητα της θάλασσας να αναπαράγει τον ηχθειοπληθυσμό της. Πρέπει λοιπόν εμείς να καλύψουμε και τις ανάγκες ε, των παρακτήων περιοχών και των νήσων. Γιατί έχει σημασία μια τέτοια πρόταση. Θα έλεγα ότι η νέα πολιτική αλληλείας, η μεταρρυθμισμένη πολιτική αλληλείας μπορεί να βοηθήσει. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ορίσουμε καλύτερα, να εξειδικεύσουμε την προσπάθειά μας στην περιοχή αυτή. Αν κάνουμε καλή δουλειά θα έλεγα στην Αδριατική μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στη Μαύρη Θάλασσα μετά που έχει αρκετά ίδια χαρακτηριστικά. Είναι μια συγκεκριμένη κλειστή θάλασσα στην οποία συμβιώνουν κοινοτικέ και μη κοινοτικέ χώρες στην οποία θα πρέπει να διασφαλιστεί η ισορροπία των δυνατοτήτων παρέμβασης, να υπάρξει μια σωστή διαχείριση των αλλιευμάτων και αυτά θα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο και με μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση, ο στόχος της πρότασης είναι αυτός. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ και αρκετές εβδομάδες, δηλαδή το είχατε στη διάθεσή σας για να το μελετήσετε. Νομίζω ότι μπορούμε να, να βάλουμε ένα όριο για την κατάθεση των τροπολογιών στις 27 του μηνός Μαρτίου και στη συνέχεια να περάσουμε στην ψηφοφορία, στην Ολομέλεια, ε, στην Επιτροπή μας μάλλον, τον μήνα Μάιο. Είμαι στη διάθεσή σας για κάποιες επιμέρους διευκρινήσεις. Να λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι αυτή στιγμή κατατέθηκε η πρόταση, έχουν μεσολαβήσει κάποια νέα δεδομένα και κάποιες επιμέρους διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν, γιατί όπως είπα έχει περάσει κάποιος χρόνος από τότε που διατυπώσαμε την έκθεση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάστακ, επόμενη στην κατάλογο μιλητών. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Μιλάνα για την έκθεσή του. Σε αυτή την περίπτωση Πρόκειται για μια στρατηγική μιας θαλάσσιας λεκάνης. Είχαμε τη στρατηγική σε σχέση με λεκάνες στην Ευρώπη. Ξεκινώ εκεί συνειδητά Ξέρετε ότι καταβάλω προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη αλληλευτική πολιτική όπου η αλληλεία διαδραματίζει ένα μεγάλο ρόλο αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος και άλλα στοιχεία επίσης. Αυτό που βρίσκω καλό σε αυτή την έκθεση είναι ότι συνδέεται η αλληλεία με την υδατοκαλλιέργεια, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε την αηφορία στην αλληλεία. Ε, ασκούνται επικρίσεις γιατί υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την αλίευση και τις αλιευτικές δραστηριότητες σε αυτή την περιοχή. Ευχόμαστε να είχαμε περισσότερα στοιχεία. Επίση υπάρχουν λίγα στοιχεία πως ο τουρισμός συνδέεται με την αλία, τι μπορεί να γίνει και είναι καλό το ότι ο εισηγητής επισημαίνει την περιφερειακή προσέγγιση, την διασυνοριακή προσέγγιση που όπως είπαμε αφορά όχι μόνο ευρωπαϊκά κράτη, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κράτη εκτός αυτής. Έχω κάποια συστήματα που με τροπολογίες θα διασφαλίσω, διότι είναι σημαντικό για μένα όχι μόνο η αηφορία στην Αλία να ληφθεί υπόψη που επί μεγάλο χρονικό διάστημα στις δραστηριότητες μας βρίσκεται στο επίκεντρο στην Επιτροπή Αλίας, αλλά για να δοθούν και κάποιες ε, προτάσεις για την θαλάσσια πολιτική, να λάβουμε υπόψη την χωροταξία στα θαλάσσια θέματα, στην, ε, ε, στα, στα θαλάσσια ζητήματα επίσης για την ολοκληρωμένη πολιτική, θαλάσσια πολιτική για τη Μεσόγειο. Είναι σημαντικό να λέμε ότι είναι σημαντικός ε, πόρος ε, για την, ε, το εισόδημα των αλλιέων η αλληλεία, όμως υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορεί να γίνουν για την αλληλεία και πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέλλον από ότι μόνο αυτό. Και επιπλέον συμβαίνει και το εξή. Πιστεύω ότι σε αυτή την πολύ μικρή αλληλή, μικρή κλίμακα βιοτεχνική αλληλεία δραστηριότητε μπορούν εξαιρετικά να συνδεθούν με τουριστικέ δραστηριότητε. Και στην Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών πολλά μπορούν να γίνουν ω προτάσει για να προαχθεί αυτό το θέμα. Όπου προσπαθούμε στην Ευρώπη να έχουμε μια στρατηγική για τον τουρισμό που θα προαχθεί, που φυσικά και τι παράκτιε περιοχέ και την αλληλεία θα λαμβάνει υπόψη θα συνδέεται με αυτήν. Πολλοί θέλουν να δουν λοιπόν αυτέ δραστηριότητε Ευχαριστώ για την έκθεση. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες και χαίρομαι για την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε κύριε Σαντινόρο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να θέσω ορισμένε ερωτήσει προ τον κύριο Μιλάνα γιατί η συνάδελφος Ματέρα η οποία είναι η σκιώδη εισηγήτριά μα, δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα και μου ζήτησε να θέσω τα ερωτήματα αυτά. και κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις ε, να προτείνω όπως είπε και ο κύριος Μιλάνα. Στην σελίδα σαν παράδειγμα 3, στην σελίδα 3 της μετάφρασης που έχω εγώ στη γλώσσα μου, ε, λες σε μία φάση ότι Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το συγκεκριμένο ταμείο, το ψήφισμα για το συγκεκριμένο ταμείο θα ψηφιστεί σύντομα. Οπότε εδώ υπάρχει ίσως κάποιο λάθος, γιατί η εντύπωση που δίνει η διατύπωση είναι ότι υπάρχει αυτό το ταμείο. Να ορίσουμε λοιπόν σωστά για ποιο ταμείο μιλάμε. Μετά από αυτό, στην επόμενη σελίδα, στην σελίδα 5, της μετάφρασης στην Ιταλική γλώσσα στο G αγγλικό, καλό θα είναι να αναφερθούμε στον αριθμό της γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών. Καλό θα είναι να έχουμε το στοιχείο, το συγκεκριμένο, του αριθμού. Πάντα στην ίδια σελίδα, στο ε, αγγλικό, θα ήθελα να καταλάβω κάτι εδώ λέει στο τέλος της παραγράφου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να ενισχυθεί με καλύτερη συνεργασία όλων των συμμετεχουσών χωρών. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ, ε, θα έλεγα, μεταφραστικό λάθος, αλλά αν ε, συμμετέχουν οι χώρες σημαίνει ότι ήδη συμπεριλαμβάνονται. Δεν ξέρω τι ακριβώς ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ. Λέτε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη ενός χωροτακτικού πλαισίου σε πολλές χώρες και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι μια έννοια με την οποία φυσικά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Από την άλλη όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το οποίο λέγεται έτσι ώστε τα προγράμματα τα οποία αφορούν την γεωργία, την θάλασσα και τον τουρισμό να οριστούν σωστά γιατί έτσι όπως προτείνεται η συγκεκριμένη διατύπωση δεν δίνει την δυνατότητα ε, σωστής κατανόησης. Ψάχνει ο μιλητής. στη σελίδα 6 λέει τώρα στο ιταλικό κείμενο λες ε, συνάδελφε ότι οι πληροφορίες που έχουμε για τους ηχθειοπληθυσμούς στη λεκάνη της Αδριατικής δεν είναι ικανοποιητική ε, η εικόνα που έχουμε. Λοιπόν, έχεις κάποιες πηγές ε, στις οποίες βασίζεσαι για να το πεις αυτό ή είναι μια φράση η οποία είναι λίγο γενικόλογη. Μετά στην παράγραφο 7. λέει ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν ως βέλτιστες πρακτικές και να επεκταθούν και σε άλλα πεδία εφαρμογής. Ποια είναι αυτά τα πεδία εφαρμογής, τι θες να πεις με αυτό. Στο σημείο 15 τώρα, λες ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με τις τρίτες χώρες, πέραν του διαλόγου που υπάρχει με τις ε, υπάρχουσες στη συγκεκριμένη περίπτωση χώρες. Πρέπει να διευκρινιστεί εδώ τι ακριβώς εννοείς διάλογο με τρίτες χώρες και στο σημείο 19 καλεί στην Επιτροπή να προτείνει τη σύσταση στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΑΚ ειδικών συμβουλευτικών οργάνων. Και ε, αναφέρεσε επίσης και στο πρόγραμμα Περιφέρειες της Θάλασσας και στις επαγγελματικές επαφές οι οποίες ισχύουν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Ε, λέει ο, ο δεν ξέρω αν περιορίζεσαι στο ΡΑΚ ή αναφέρεσαι και σε άλλου είδους επαγγελματικές οργανώσεις. Ευχαριστούμε η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλάνα. Θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε αυστηρά λιευτικά θέματα. Και θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις, κυρίως ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Όταν εσείς λέτε στο σημείο 12 ότι στην λεκάνη του Ιωνίου και της Ιαδριατικής υπάρχει ένα είδος αλλιευμάτων που απαιτεί ξεχωριστής ε, μορφής αλλιεία και ένα ενιαίο πρόγραμμα διαχείρισης. Πώς το δικαιολογείτε αυτό διότι θυμάμαι ότι είχαμε κατά το παρελθόν όταν είχαμε μια πρόταση που από την Επίτροπο Μπονίνο απέρευσε για την μείωση του ελάχιστου μεγέθους ε, για το Μερλούκιο στην Αδριατική καταλήξαμε τότε στο συμπέρασμα και αυτό ήταν πρόταση για το, τα αλλιεύματα όπως και αλλού στη Μεσόγειο ότι δεν είχε κανένα νόημα η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ε, δικαιολογεί το το μόνο πρόβλημα ήταν ότι αλίευαν σε κάποιες ζώνες γόνων και έτσι ε, συλλάμβαναν τα μικρότερα ψάρια, αλλά όχι πρόγραμμα ξεχωριστής διαχείρισης. Ε, με λοιπόν, σε τι βασίζετε εσείς στο επιχείρημά σας ότι χρειάζεται ένα ξεχωριστό σχέδιο διαχείρισης για αυτή τη ζώνη, όταν εγώ έχω πληροφορίες ότι δεν δικαιολογείται αυτό, διότι είναι πολύ ευρύτερο το αλίευμα από ότι στην λεκάνη της Αδριατικής ε, και του Ιωνίου. Δεύτερη παρατήρηση, Όσο αφορά το στο σημείο 14. Όταν γίνεται πρόταση κανονισμού για τεχνικά μέτρα για την ζώνη του Ιωνίου και της Αδριατικής και γι' αυτό θα ήθελα το θέμα αυτό να γνωρίζω ποιο είναι το σκεπτικό το οποίο, στο οποίο βασίζεστε. Δεν κατανοώ γιατί στην Μεσόγειο πρέπει να υπάρχουν τμήματα με διαφορετικού είδους διαχείριση και μέτρα από ό,τι σε άλλα. Και όταν έχουμε το θέμα του Συμβουλίου Αλλιέας για τη Μεσόγειο, που ακριβώς καταβάλει προσπάθεια βήμα προς βήμα για να καταλήξουμε σε κοινά τεχνικά μέτρα για όλη τη Μεσόγειο και για όλες τις χώρες ε, της Μεσογείου, είτε είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, θεωρώ ότι αυτή η διαφορετική πρόταση εδώ δεν έχει μεγάλο νόημα, αυτή η διαφοροποίηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται αυτό, δεν, δεν τεκμηριώνεται. Δεν... Εσείς μπορείτε να μου αποδείξετε το αντίθετο, ότι χρειάζεται και να με πείσετε. Και για το επόμενο θέμα, το 15 με το οποίο συνδέεται αυτό το θέμα, η σχέση με άλλες χώρες ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνεται μέσω των περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτές οι περιφερειακές οργανώσεις πρέπει πολύ περισσότερο να ενισχυθούν. Είναι όμως ε, μέσω του ERP ε, της περιφερειακής οργάνωσης αλίας μέσα στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να συμφωνούνται τα τεχνικά μέτρα τα οποία θα ισχύουν και πρέπει να ισχύουν για όλη τη Μεσόγειο. Αυτά είναι τα γενικά μου σχόλια. Εκτός αν εσείς αποδείξετε ότι αυτά που λέτε είναι σωστότερα και σε αυτή την περίπτωση θα υποστηρίξω την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γαρθία Γέρο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μιλάνα, τον συνάδελφό μας και φίλο Μιλάνα για το έργο που επετέλεσε, διότι ήταν σημαντική επιτυχία σε αυτό το θέμα και με την επίσκεψη που κάναμε ως αποστολή με αυτή την περιοχή και το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Σήμερα συζητάμε αυτό το θέμα σχεδίου έκθεσης για το, την Αδριατική και το Ιόνιο και πέρασε λίγος χρόνος, λίγοι μήνες από τότε και προχωράμε και προσπαθούμε η κοινοβουλευτική μας επιτροπή, οι συντονιστές να λάβουν υπόψη το σχέδιο της έκθεσης για τη συνεισφορά των γυναικών στον αλλιευτικό τομέα στην Ευρώπη. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί όμως τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σε εσάς. Δεν ασκώ επικρίσεις, ε, όμως το θέτω αυτό ως θέμα όταν συμβαίνει καμιά φορά πράγμα, κάτι τέτοιο όταν είναι κάποιος ε, ε, άπειρος ή νεότερος ε, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη αυτά σε σχέση με το παρελθόν. Θέλω να σας συγχαρώ εν πάση περιπτώσει για την παρουσίαση και την αναφορά που πρέπει να γίνει σε δύο θέματα και που θεωρώ ότι δεν είναι αντιφατικά ή θα ήθελα να μου το αποσαφηνίσετε να ενταχθεί ο ρόλος που πραγματικά έχουν οι γυναίκες σε αυτόν τον τομέα, στην ανάπτυξη, στην αλία και η οικονομική συνεισφορά από πλευρά του, διότι βρισκόμαστε σε δύσκολε οικονομικές περιόδους, σε δύσκολη συγκυρία και για τις ε, γυναίκες ε, και την ανεργία και που πλήττονται από αυτήν Πρέπει να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε την κατάρτισή τους και την δυνατότητα συμμετοχής τους ε, στην εργασία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κατά ποιο τρόπο δικαιολογείται από πλευρά σας ε, ότι γίνεται εδώ λόγος ε, για την υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας. Θα ρυθμιστεί σε σχέση με το PPC, καθώς επίσης και τη διάθεση στην αγορά μέσω των κοινών οργανώσεων αγοράς και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα από πλευράς ταμείου. Για να μην επεκταθώ υπερβολικά θέλω να πω ότι ανησυχώ για το πώς μπορεί να επιληθεί το ζήτημα. Ότι πραγματικά μέσα σε μια στρατηγική για τη Μεσόγειο θάλασσα θα πρέπει να δούμε δυνατότητα ε, κάποιου, κάποιας πρόσθετης αξίας που μπορεί να δημιουργηθεί. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο θέμα που είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση που στο τέλος τέλος όταν θα έχουμε ευκαιρίες να επικεντρωθούμε σε αυτά θα πρέπει να δούμε τροποποιήσεις ε, προτάσεων Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε και να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τις τρίτες χώρες, όπως ε, για παράδειγμα στην περιοχή της Μεσογείου. Και επ' αυτού θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και για κάτι το οποίο λειτουργεί, πώς είναι δυνατόν κάτι να ε, πρέπει πάλι να αλλάξει και να μην μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ένα μόνο και τελευταίο θέμα που αφορά την εργασία μας εδώ. Ο πρόεδρος ε, που σε πολλά θέματα που ε, είδαμε σήμερα έχει δίκιο. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε εδώ αποφάσεις έχουν, ε, όταν έχουν συζητηθεί αυτά τα πράγματα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και έχουν το προηγούμενο βράδυ μόνο διατεθεί μεταφράσεις ε, στα ισπανικά. Το, ε, αρνούμε να εργαστούμε με, άλλη, με άλλο τρόπο, να τροποποιήσουμε τον κανονισμό μας και τη συνθήκη της Λισαβόνας και να εργαζόμαστε με τρόπο που δεν είναι αποτελεσματικός. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις και προτού δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μιλάνα, η Επιτροπή. Θα ήθελε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μελάνε για αυτή την έκθεση, την οποία καλωσορίζει η Επιτροπή. Όπως σας είπα και στην τελευταία μας συνάντηση. Όταν συζητήθηκε αυτή η έκθεση, θεωρούμε ότι είναι κέρια και ταιριάζει με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και η Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ε, κοινή πολιτικής αλίας. Και αυτή η πρόταση για να πάμε περισσότερο προς την περιφερειακή ε, διαχείριση της αλίας που μπορεί να εφαρμοστεί ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περιοχή του Ιωνίου για της Ιαδεατρικής. Το Δεκέμβριο του 2012 υιοθετεί η Επιτροπή μια ανακοίνωση για την στρατηγική της θαλάσσιας αλίας στην Αδριατική και το Ιόνιο, με το οποίο προτείνεται ένα πλαίσιο δράσης και ένα σχέδιο δράσης για το 2013. Εν τω μεταξύ υπήρξαν εξελίξεις που πιθανώς θα τις γνωρίζετε. Μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ανατέθηκε στην Επιτροπή η δημιουργία μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Αδριατική και το Αιώνιο σε συνεργασία με τη Γενική ε, Διεύθυνση Αλίας θα εργαστούμε για την κατάρτιση αυτής της στρατηγικής και ενός ε, πλήρους σχεδίου δράσης το οποίο θα υλοποιηθεί το 2014. Αυτό το κοινό και ενιαίο σχέδιο δράσης θα έχει μια ενότητα που θα αφορά τις ε, δράσεις για την ε, θάλασσα, ιδίως για ε, την αλία και την υδατοκαλλιέργεια. Και θεωρώ λοιπόν ότι πολλές από τις προτάσεις σας μπορούν να συμπεριληφθούν εκεί, σε αυτό το σχέδιο δράσης. Προφανώς οι χώρες της Αδριατικής ε, θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να αποφασίσουν ποιες δράσεις θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο. Θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία συνεργασίας με, αυτή της, με τις χώρες αυτής της περιοχής για να εξευρεθούν τα πιο κατάλληλα και χρήσιμα ε, προγράμματα προς την κατεύθυνση που έχετε περιγράψει και στην εκθεσή σας. Θέλω τώρα σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα να αναφερθώ. Και να αναφερθώ και σε αυτά που είπαν και κάποιοι προλαλήσοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το πλαίσιο της, ε, του κανονισμού για τη Μεσόγειο, για την αλία στη Μεσόγειο, που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του βυθού στη Μεσόγειο, της ε, λεκάνης της Μεσογείου, καθώς επίσης και τις ε, υποπεριφερειακές στρατηγικές, με την υιοθέτηση σχεδίων διαχείρισης, τα οποία εγκρίνονται είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει πάλι η δυνατότητα αυτά τα σχέδια διαχείρισης να εγκρίνονται σε, ε, μεταξύ πολλών κρατών, σε διεθνικό επίπεδο. δεν βλέπουμε το λόγο να υπάρξει μια συγκεκριμένη ξεχωριστή, ε, κανονισμός ειδικά για την ιατρική για τον Ιόνιο, γιατί η γενικότερη κατεύθυνση της περιφερειακής στρατηγικής για την Αλία θα μας δώσει τη δυνατότητα να την εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική και σε πιο συγκεκριμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα η ιατρική. Συμφωνούμε μαζί σας ότι στην λεκάνη της Αδριατικής και του Ιουνίου πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι βρίσκονται και χώρες που δεν είναι ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιούνιο και η Κροατία, αλλά και τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν, τα θέματα του Ιωνίου και της Αδριατικής θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της Γενικής Επιτροπής για την ε, Αδριατική. που έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αναθεώρησης στην οποία ε, δραστηριοποιείται έντονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή συγκεκριμένα. Ξετάζουμε την πιθανότητα να προταθεί ένα πολιετές σχέδιο διαχείρισης αλλιευμάτων. Θα υποβάλουμε τη σχετική πρόταση στην Γενική Συνέλευση του Μαΐου συνεργαζόμαστε στο τεχνικό επίπεδο και μόλις είμαστε σε θέση να υποβάλουμε τη σχετική πρόταση θα σας ενημερώσουμε και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή σας ε, να γνωμοδοτήσει. Υποβάλλοντας τη σχετική πρόταση. και προφανώς ε, ευελπιστούμε να συνεργαστούμε μαζί σα σε αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Μιλάνα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ όλου για την προσοχή που δώσατε στην πρόταση. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το ενδιαφέρον αυτό και από τη συζήτηση που προηγήθηκε, που θα οδηγήσει σε βελτιώσεις θα προσπαθήσω να ακολουθήσω μια κάποια σειρά, αν τυχόν κάτι μου διαφύγει θα επανέλθω. Θα αρχίσω από τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Σαντινόρο. Λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, εκεί που υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης θα γίνει. Για τις ε, λιγότερο τυπικές και πιο ουσιαστικές θα έλεγα παρεμβάσεις, Ξεκινάω από το O αγγλικά. Στη σελίδα 6 του Ιταλικού κειμένου. Υπάρχει το θέμα της χωροταξίας εδώ το οποίο τίθεται. Θα ήθελα να πω ότι γενικά υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά πρόσφατη Δεν ξέρω αν υπάρχει λοιπόν εδώ δυνατότητα σύνδεσης με τον συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο ο οποίος μας απασχολεί. Όλες οι μορφές χωροταξίας έτσι όπως ασκείται και σχεδιάζεται εν πάση στην Ευρώπη στην ουσία δεν έχουν οδηγήσει πουθενά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα δεν είναι να πούμε ποια περιοχή είναι οικοδομήσιμη και ποια δεν είναι οικοδομήσιμη. Απλά θα πρέπει να ορίσουμε σε επίπεδο περιφερειακό ποιες είναι οι συνθήκες που θα πρέπει να κρατούν στην περιοχή και πώς θα πρέπει να προκρίνουμε κάποιες δραστηριότητες ε, και όχι κάποιες άλλες. Οι θαλάσσιες περιοχές γενικά δεν έχουν γίνει αντικείμενο προγραμματισμού. Όλα γίνονται αθόρμητα θα έλεγα και πολλές φορές υπάρχει μια κάποια σύγχυση και κάποιες αντιφατικές καταστάσεις στις παράκτιες περιοχές όπου περιοχές αλληλείας έρχονται σε σύγκρουση με περιοχές υδατοκαλλιεργιών, με περιοχές τουριστικές, με αστικές περιοχές κτλ. Το θέμα είναι γενικότερα για την Ευρώπη ε, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της χωροταξίας πέραν της ακτής να συμπεριλάβουμε και την ε, θάλασσα στην αντίληψη που έχουμε <clears throat> για την χωροταξία και τις χωροτακτικές ρυθμίσεις. Εγώ θέλησα λοιπόν να εισάγω το συγκεκριμένο στοιχείο και να το θέσω στην ε, ε, προσοχή σας έτσι ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να επηρεάσουμε και την ολοκληρωμένη αλλιευτική πολιτική σε αυτή τη λεκάνη. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πιλωτική δράση κατά κάποιο τρόπο και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα και προς την χωροτεκτική αυτή ε, πρακτική. Υπάρχουν ε, όλοι οι παράγοντες οι οποίοι παίζουν κάποιο ρόλο μεταξύ των οποίων και οι σχέσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες και μη ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία περιοχή στα πλαίσια της οποίας οι χωροτακτικές ρυθμίσεις μπορούν έστω και σε πειραματικό επίπεδο να ε, εφαρμοστούν προκαταλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο το τι μπορεί να ακολουθήσει στην Ευρώπη γενικότερα. Όπως είπα λίγο πριν, από τότε που γράψαμε το κείμενο μέχρι σήμερα έχουμε μεσολαβήσει διάφορα και αυτά θα προσπαθήσει να τα διορθώσουμε. Το είπε και η εκπρόσωπος, τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε η πρόταση της Επιτροπής για τη χωροταξία, υπήρξε η πρόταση για τη στρατηγική εντωμεταξύ της Αδριατική που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ειδικέ προτάσεις για το σύνολο της περιοχής ευρύτερα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία φάση θα έλεγα ανωδική δημιουργίας κανόνων και ρυθμίσεων. Θα πρέπει όμως να παρέμβουμε άμεσα και στον τομέα της θάλασσας έτσι ώστε η αλληλεία να μην θεωρηθεί ο φτωχός συγγενής των υπολείπων συμφερόντων και δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι βιώνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή σε σχέση με τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Χωρικός προγραμματισμός λοιπόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις οικονομικές δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάποιες περιοχές θαλάσσιες σημεί θα έλεγα και ε, μέσω ανάπτυξης και μέσω παροχής εγγυήσεων για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων. Τώρα για τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Είναι σαφές ότι αυτά τα οποία είπαμε προβλέπονται αλλά δεν γίνονται. Προβλέπονται διμερείς σχέσεις με τις χώρες αυτές αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Οκτώ κοινοτικέ χώρες, 14 μη κοινοτικέ χώρες. Οκτώ χώρες οι οποίες είναι υποχρεωμένες λόγω των κανονισμών να σέβονται κανόνες αυστηρούς, ε, αυστηρούς για ε, την αλληλεία, για την αλληλευτική δραστηριότητα και 14 χώρες οι οποίες σκοτίστηκαν για αυτούς τους ε, αυστηρούς κανόνες. Σε σχέση λοιπόν με την ανυπαρξία των σημερινών σχέσεων θα πρέπει και στα πλαίσια της Επιτροπής και στα πλαίσια των επιμέρους υποεπιτροπών και στα πλαίσια των ΡΑΚ να παραδεχθούμε ότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Καμία χώρα μεσογειακή μη κοινοτική δεν εφαρμόζει τους κανόνες που εμείς σεβόμαστε και εφαρμόζουμε. Γιατί λοιπόν μιλάμε για μια συγκεκριμένη ε, μικρή θαλάσσια περιοχή, κλειστή θαλάσσια περιοχή και ο ανταγωνισμός ας πούμε ανάμεσα στην Κροατία και τη Σλοβενία, δεν θέλω να αναφερθώ, είναι κάτι το θα έλεγα δολοφονικό γιατί στην ουσία βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους και μέσα σε συγκεκριμένες μικρές θαλάσσιες ζώνες σε κάποια σκάφη σέβονται τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς και κάποια άλλα κάνουν ό,τι θέλουν και σε επίπεδο ανταγωνισμού και σε επίπεδο συνθήκων γενικότερα. Το είδατε και στη Βενετία όταν είχατε έρθει ότι υφιστάμεθα πραγματικά συνεχώς ε, ε, επιθέσεις ουσιαστικά από ε, τους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν εδώ να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια έκτακτη προσπάθεια η οποία να διαφεύγει θα έλεγα από τις κανονικές διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων οριμάζουν οι διεθνείς σχέσεις. Ε, μια έκτακτη προσπάθεια λοιπόν στα πλαίσια της οποίας να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση ανάμεσα στις κοινοτικές και μη κοινοτικές χώρες που να εφαρμόζουν τουλάχιστον τους ίδιους κοινούς κανόνες. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια στην εφαρμογή αυτής της ε, αρχής, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως παρόλα αυτά εμείς καλούμεθα Ιταλία, Σλοβενία και σιγά σιγά και Κροατία να συνεννοηθούμε. Οι υπόλοιποι κάνουν ό,τι θέλουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί σεβόμεθα διαφορετικούς κανόνες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ειδική προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό που είπα ανταποκρίνεται σε αρκετές ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις της κυρίας Φράγκα, πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω και εγώ σε σχέση με αυτές. Η Αδριατική αντίθετα από όλη την υπόλοιπη Μεσόγειο. Είναι μια διαφορετική θάλασσα. Στο Τυρινικό πέλαγο, σαν παράδειγμα, και αναφέρομαι στην Ιταλία. Γιατί Ιταλός είμαι, αυτά ξέρω. Στο Τυρινικό πέλαγος έχουμε κάποιες ε, πλάκες, θα έλεγα, 30-40 μέτρων βάθος, στα 30, 40 ή 50 μέτρα από την ακτή. όλο το τυρινικό πέλαγος είναι φτιαγμένο έτσι. Στην Αδριατική για να φτάσεις στα 50 μέτρα πρέπει να φύγεις 50 μίλια από την ακτή. Στο ένα μίλι είσαι στα 3 μέτρα, στα 3 μίλια είσαι στα 10 μέτρα βάθος. Έχουμε λοιπόν ε, κανόνες σε επίπεδο Μεσογείου που επιβάλλουν μία απόσταση από την ακτή και δεν υπάρχουν δυνατότητες παρεκκλήσεων και εξαιρέσεων. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν απαιτείται η τροποποίηση του κανονισμού και απαιτείται αυτές οι συνθήκες οι διαφορετικές που ισχύουν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν. Υπάρχουν λοιπόν και ορισμένες αλλιευτικές δραστηριότητες, τις είδαμε στη Βενετία. Είδαμε ότι απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές και αλλιεύσεις όριμων ηλικιακά πληθυσμών. Υπάρχει ένα μικρό αλλιεύμα στη συγκεκριμένη περιοχή του οποίου ε, απαγορεύεται εν πάση περιπτώσει η αλλιεία σε αυτή τη φάση. θα μπορούσα να αναφερθώ σε 7 ή 8 επιμέρους ρυθμίσεις που δεν είναι εφαρμόσιμες στην Αδριατική ή που εν πάση περιπτώσει υπονομεύουν τις αλλιευτικές δραστηριότητε και δεν είναι καθόλου χρήσιμες σε επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος και πρέπει να τροποποιηθούν. Δεν μπορώ φυσικά σε αυτή την έκθεση που είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας να ορίσω συγκεκριμένα όλες αυτές τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά και από πλευρά των επαγγελματικών οργανώσεων και από πλευρά των οργανώσεων των αλλιέων και από πλευρά των ΜΚΟ προστασία του περιβάλλοντος. Ζητείτε ορισμένοι κανόνες στην Αδριατική να αλλάξουν γιατί δεν είναι εφαρμόσιμοι. Υπάρχουν λοιπόν όχι μόνο αντιφάσεις στο εσωτερικό των κανονισμών αλλά ανάγκες για καλύτερες διευκρινήσεις. Από την ανάλυση λοιπόν την οποία θα κάνουμε θα μπορέσουμε ίσως ε, να βρούμε λύσεις, αλλά λύσεις δεν βρίσκονται στα πλαίσια των διαχειριστικών προγραμμάτων λόγω της μορφολογίας που παρουσιάζει η Αδριατική. Νομίζω ότι απάντησα σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Στα πλαίσια της χωροταξίας υπάρχει η ευρύτερη ένταξη στην ε, μεσογειακή πολιτική και στην συνεργασία της αλλιευτικής δραστηριότητας με τις τουριστικές δραστηριότητες. Και για τις τρίτες χώρες μίλησα και για τα ΡΑΚ μίλησα Τώρα για το ειδικό ρακ που έθεσε ο Αντινόρο, όχι δεν θέλουμε ένα ειδικό ρακ. Λέμε ότι στα πλαίσια μια καλύτερα διευκρινισμένης στρατηγικής, το ρακ για την Αδριατική, να έχει περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας. Να έχει κάποια ειδικότερα εδαφικά χαρακτηριστικά. Εγώ δεν λέω ότι λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Όχι, πρέπει να είναι μία η πολιτική η μεσογειακή. όλα αυτά, στο εσωτερικό αυτών των θαλασσίων περιοχών υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τίθενται με διαφορετικό τρόπο και πρέπει να συζητηθούν πιο εξειδικευμένα. Όλοι οι οργανισμοί στους οποίους αναφερθήκατε, και εγώ επιμένω σε αυτό, δεν επηρεάζουν τελικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί δεν έχουν βρει λύσεις στα θέματα τα που αφορούν σαν παράδειγμα την περιοχή ανάμεσα στην την Ισία, τη Λιβύη και τη Σικελία. Και μετά από την ε, Άνοιξη την Αραβική και την Επανάσταση αναφερθήκαμε θα έλεγα στην αλαζονία ορισμένων χωρών ή ορισμένων διεθνών οργανισμών δεν οδηγηθήκαμε πουθενά. Δεν υπήρξε κανένα μα κανένα θέμα το οποίο να λύθηκε με συντονισμό στον τομέα σαν παράδειγμα των ελέγχων. Πώς θα ελέγξουμε τη Μεσόγειο. Και η υπηρεσία του Βίγκο με τις δορυφορικές δυνατότητες που έχει κάνει λίγα πράγματα. Αλλά όταν έχουμε από τη μία οκτώ κοινοτικέ χώρες και από την άλλη 14 μη κοινοτικέ. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι διεθνείς οργανισμοί αφήνουν ε, κάθε ελευθερία σε όσους ασκούν δραστηριότητε στις περιοχές. Ξέρουμε τι γίνεται και στον τομέα του τόνου στη Μεσόγειο και σε σχέση με τις δυνατότητες σεβασμού των ποσοστώσεων που έχουν προκαθοριστεί. Ξέρουμε ποιες είναι οι παράνομες δραστηριότητες. Ξέρω επίσης ότι το να τα λέω αυτά τα πράγματα εδώ δημιουργώ άσχημο κλίμα, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς υπάρχουν 14 μη κοινοτικέ χώρες. και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με ενιαίο τρόπο Ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιοχές κλειστές όπως η Μαύρη Θάλασσα η οποία έχει ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη Μεσόγειο και μπορεί να κάνει επιμέρους ειδικέ ρυθμίσεις. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να εμβαθύνω λίγο σε κάποιες από τις σκέψεις τις οποίες εκφράσατε. Δεν σας κρύβω ότι επειδή ακριβώς τους τελευταίους μήνες έχουν τροποποιηθεί ορισμένα στοιχεία και έχουν υπάρξει ορισμένα καινοτόμα στοιχεία, το κείμενο είναι τροπολογήσιμο και θα ήμουν ιδιαίτερος ευτυχής αν καταθέσετε τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Θέλατε να λάβετε τον λόγο. Εντάξει και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ σε επίμαχα θέματα και να κάνουμε κάποια πολεμική εδώ, αλλά θα ήθελα να προσαφινιστεί ένα πράγμα. Ας το δούμε αυτό. Για τη Μεσόγειο και για το σύνολο της Μεσογείου. Αναφέρομαι στους αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια απόρριψη όσον αφορά τον κανονισμό τεχνικών μέτρων. Απόρριψη από πλευρά τους. Απόρριψη που σε κάποιο σημείο μπορεί να δικαιολογείται ή όχι. Όμως ευθύ εξ αρχή απόρριψη. Είμαι εισηγήτρια για αυτό το θέμα και ξέρω τι σήμαινε για να προχωρήσει αυτός ο κανονισμός σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά καλά αυτό το θέμα, διότι με αυτή την αφορμή είχα την δυνατότητα να συναντήσω όλους του τομέα αυτού. Τώρα, όταν λέγεται ότι αυτός ο κανονισμός έχει ένα σκεπτικό σε σχέση με το που μπορεί να αλλιεύει κανείς σε σχέση με την ακτή και την απόσταση από την ακτή που ήταν ένα από τα πιο επίμαχα θέματα, γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά για ποιο πράγμα γίνεται λόγος εδώ, σε αυτό το θέμα υπήρχε μεγάλη ελαστικότητα και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κριτηρίων μέσω των οποίων μπορεί να τροποποιείται όταν δικαιολογείται τεχνικά και ε, επιστημονικά το θέμα σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Μια και όλο το όλη η Μεσόγειος δεν είναι παρόμοια και σε σχέση με την απόσταση υπάρχουν θέματα που πρέπει να διαφοροποιούνται. Αυτό αρκετά καλά αποσαφηνίζεται στον κανονισμό και νομίζω ότι δεν είναι αποδεκτή η επίκριση που ασκείται από πολλούς αληθεύει ότι σε κάποια στιγμή θα έπρεπε να, σε σχέση με σχέδια και την κατάθεση, κατάθεσή τους, όμως όταν λέγεται ότι ο κανονισμός αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και που είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη και όταν ακούγονται αυτά ως επικρίσεις, αφενός αυτό από την άλλη Συνεχίζω να εμένω και να επιμένω ότι όταν κάνουμε μ, κανονισμούς για κάποιες ε, ζώνες ε, και όταν υπάρχει το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, όταν λέμε ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν κάποια πράγματα για τη Μεσόγειο, θα μπορούσαν να βελτιωθούν ιδιαίτερα όσον αφορά το μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων που υπάρχουν για αυτόν τον κανονισμό, για τις πιέσεις που ασκούνται από πλευράς ε, ε όσων εμπλεκόντουσαν στον τομέα αυτό. Αυτό αφενός. Από την άλλη πλευρά, να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί με αυτόν τον κανονισμό. Και θα ήθελα να πω ότι όλα εντάξει μπορούν να βελτιωθούν. Αλλά η λύση δεν είναι να έχουμε 20 κανονισμού τεχνικών μέτρων για την περιοχή της Μεσογείου. Δεν συμφωνώ με μια τέτοια τοποθέτηση. Και μετά δράτω με τις ευκαιρίες, Πρόεδρε, για το θέμα που αναφερθήκατε για τον ε, και, ε, ε τόνο σε σχέση με τους ε, υπεύθυνου για την κατάσταση αυτή. Και εδώ σε σχέση με εμάς λέγαμε ότι το πλεονάζον δυναμικό που υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεία αυτού του είδους δεν μπορούμε να ρίξουμε το φταίξιμο σε όλους αδιάκριτα. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν τα πράγματα και υπήρξαν προσπάθειες, γι' αυτό βελτιώθηκε η κατάσταση του κιανόπτερου τόνου και κάναμε προσπάθειες και κάποια στιγμή ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούμε να δώσουμε στοιχεία σε σχέση με τους ε, στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτούς τους λόγους τώρα υπήρξε ρύθμιση του τομέα και ανέκαμψε το αλίευμα. Και πράγματι βελτιώθηκε το απόθεμα, το, το αλίευμα του κυανόπτερου τόνου. Πρέπει να δούμε ότι και σε, ε, σχέση με άλλες χώρες ε, επειδή έλεγαν ότι είναι η κύρια υπεύθυνη Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είχε τη μεγαλύτερη ποσόστοση λοιπόν σε σχέση με τρίτες χώρες πολύ ωραία να, αναφερθούν αυτά αλλά πρέπει να επιληθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σε σχέση με τη Μεσόγειο η Μεσόγειο είναι η μόνη ζώνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπάρχουν ούτε τάξα ανώτατα επιτρεπόμενα αλλιεύματα ούτε ποσοστώσεις και θα ήθελα να πω ότι όλα τα να με το ίδιο μέτρο και να ισοπεδώνουμε. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έγινε και για τη Μεσόγειο έγιναν πολλά πράγματα. Είναι λιγότερο ε, ε, υποκαθεστώς ρύθμισης σε σχέση με τις ζώνες αυτές και πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν τις ευθύνες τους. Είναι καλύτερο να έχουμε ένα κανονισμό τεχνικών μέτρων τον καλύτερο δυνατό που μπορούμε να πετύχουμε και δεν επιλύονται τα προβλήματα με το να έχουμε πολλούς διαφορετικούς κανονισμούς τεχνικών μέτρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε εσείς τον λόγο για να ολοκληρώσουμε παρακαλώ. Ε, Μα θα συμφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να τα κάνει από κοινού αυτά που μπορεί να κάνει. Τα υπόλοιπα δεν μπορεί να τα κάνει και εκεί είμαστε αδύναμοι. Γνωρίζω σαν παράδειγμα στην Ιταλία Ε, περάσαμε από 60 σκάφη για τον ερυθροπτέρυγο τόνο στα 16 αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω λοιπόν ότι ε, διαπιστώνουμε πια ότι το είδος αυτό έχει συγκεκριμένους μηχανισμούς άμυνας και με τα μέτρα τα οποία παίρνουμε μπορούμε να βοηθήσουμε σε μια πιο γρήγορη ανάκαμψη η Ένωση δεν είναι, η Ένωση δεν είναι να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχει ή δεν έχει τώρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή η οποία είναι κλειστή, έχουμε να κάνουμε με μια λεκάνη στην οποία συνυπάρχουν 8 κοινοτικέ χώρες και 14 μη κοινοτικέ χώρες. Και το σύστημα επικοινωνίας που έχουμε και οι οργανισμοί που έχουμε στα πλαίσια των διεθνών μας σχέσεων αποδεικνύονται συστηματικά ανεπαρκείς. Όταν κάνω καταγγελίες ε, για ε, σκάφη τα οποία ε, αλλιεύουν τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο από τις ποσοστώσεις τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους, δεν αναφέρομαι στα κοινοτικά σκάφη, αναφέρομαι στις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σαφής επιτάχυνση των πολιτικών παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Αγαπητή Κάρμεν, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σου στα υπόλοιπα και για τον κανονισμό. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος σίγουρα κανονισμός, ο οποίος όμως να έχει αρκετές δυνατότητες να εφαρμόζεται με τρόπους αντίστοιχους με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Υπάρχουν λοιπόν σε ορισμένες περιπτώσεις ανάγκες για διαφορετικά όρια. Σαν παράδειγμα, έχουμε σε μια περιοχή σχετικά περιορισμένη της Ιταλίας, ε, στην περιοχή της Λιγουρίας, συγκεκριμένες ε, ε, ρυθμίσεις, ρυθμίσεις οι οποίες έχουν δώσει ευεργετικά αποτελέσματα, οι οποίες όμως δεν ισχύουν λίγα μέτρα δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εγώ επανειλημμένα έχω προσπαθήσει να εξηγήσω στις αρμόδιες αρχές ότι οι ρυθμίσεις αυτές, ας πούμε 15 χιλιόμετρα από την ακτή στη Λιγουρία, απαγορεύουν ουσιαστικά σε μια μεγάλη κατηγορία αλλιέων να ασκούν τη δραστηριότητά τους. Εγώ δεν θέλω να έχουμε, θα έλεγα, τη Μάγνα Κάρτα ή τις 10 εντολές. Δεν είναι εκεί το θέμα για τη Μαύρη Θάλασσα ή για την Αδιατική. Το θέμα είναι ότι ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιοχή όταν αυτό χρειάζεται. Και αν σε μία περιοχή απαιτείται ένα διαχειριστικό πλαίσιο διαφορετικό με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί όχι. Θα συζητήσουμε αύριο την έκθεση του, του κυρίου Αρσένη για την αλληλεία σε μεγάλα βάθη. Ε, θα δούμε στα πλαίσια της συζήτησης αυτής τον τρόπο με τον οποίο θα θέσουμε ε, το θέμα κάποιων συγκεκριμένων αυστηρών τεχνικών ρυθμίσεων. Και φοβούμεθα φυσικά ότι οι επιπτώσεις από τα νέα αυτά μέτρα θα είναι ιδιαίτερα αρνητικά για τους αλείς και αυτοί οι οποίοι φοβούνται για τις κοινωνικο-οικονομικές ε, επιπτώσεις έχουν δίκιο. Κανένας όμως δεν έχει σκεφτεί αυτά ειδικά για την Μεσόγειο. Ο Αντινόρο γνωρίζει πολύ καλά το θέμα όπως και εγώ και έχει πάει και έχει συζητήσει με τους αλληλείς στην Αδριατική και έχει εκπλαγεί θα λέγαμε σε σχέση με τις ε, ιδέες τις οποίες είχαμε. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι οι κανόνες υπάρχουν, αλλά δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι οι δέκα εντολές. Είναι κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να τίθενται υπό συζήτηση, υπό αμφισβήτηση αν αυτό χρειάζεται και να υπάρχουν αλλαγές αν αυτό χρειάζεται να επαληθεύεται επίσης το στάδιο εφαρμογής των τεχνικών αυτών ρυθμίσεων. Εγώ λοιπόν λέγω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την δυνατότητα και επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάμε για νομοθετική πρόταση αλλά μιλάμε για συμβουλευτική πρόταση να ληφθούν ορισμένα πράγματα υπόψη, να ονοματιστούν ορισμένα πράγματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε για λόγους συνοχής στην ουσία ε, θα μείνουμε στην επιδερμική εξέταση των πραγμάτων. Ε, δεν έχει νόημα. Εμείς για να νομοθετήσουμε θα πρέπει να μπούμε στην ουσία, θα πρέπει να βυθιστούμε στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. ώρα παρακαλώ. Ε, Κοιτάξτε, δεν θέλω να, να και θα θέλω να μ' ακούσει η Κάρμεν. Σε ακούω, λέει η Κάρμεν. Κοιτάξτε, και εγώ θα μπορούσα μιλώντας να προχωρήσω σε ακαδημαϊκές παρεμβάσεις, όχι επειδή είμαι Ιταλός, αλλά γιατί προσπαθώ να ακολουθήσω τη λογική. Μένω σε αυτό που έμενε η Κάβεν Φράγκα, ότι πρέπει να υπάρξει ενιαίος κανονισμός. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ενιαίος κανονισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κάτι το θετικό. Δεν θέλω να δίνουμε μάχες άχρηστες μεταξύ μας, αλλά θα έλεγα, όπως ακριβώς το είπε και ο κύριος Μιλάνα, στην έκθεση πρωτοβουλίας του, η οποία έχει τη συγκεκριμένη αξία που έχει. Δεν είναι νομοθετική πρόταση, αλλά παρόλα αυτά κάποιες από τις αποκλήσει υπάρχουν, όχι για να κάνουν οι διάφορες χώρες ό,τι τους περνάει από το κεφάλι, αλλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να συμβιώσουμε, γιατί υπάρχουν χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι και η Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων θα ασχολείται με αυτά τα οποία ασχολείται σημαντικά πράγματα, αλλά και με το θέμα της γειτονίας, με τις χώρες της Όμορες, γιατί εκεί έχουμε θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι ένας κανονισμός πιο συγκεκριμένος θα μας επιτρέψει να περάσουμε στην απλή επιβίωση των αλλιέων μας γιατί πέραν αυτού δεν φανταζόμαστε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη παρέμβαση, καμία άλλη. Πολύ καλά. Ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο. Και να αναφέρω ότι η κατάθεση τροπολογιών εκπνέει στις 27 Μαρτίου. 27 το μεσημέρι, 12.00. Περνάμε στο επόμενο σημείο. 11. Τροποποίηση κανονισμού 1224 Συμβουλίου με θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την διασφάλιση της τήρησης κανόνων κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Αυτό το θέμα ήδη το θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και έτσι θα δώσω τον λόγο πρώτα στην Επιτροπή για να παρουσιάσει τις προτάσεις της. Αν συμφωνείτε, ο κύριος Πένας λοιπόν, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η πρόταση που μας φέρνει εδώ σήμερα είναι μια πρόταση από κοινού με άλλες που εξετάσατε προηγούμενα σε προηγούμενους μήνες προσαρμογής του κανονισμού συστήματος ελέγχου συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν είναι μια πρόταση που στόχο έχει να προσαρμόσει στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, της κατεξουσιοδότηση πράκτης, πράξης ε, και της κατεντολήν πράξης. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό ευθύ εξ αρχής. Να το πούμε δεν υπάρχει καμιά αλλαγή επί της ουσίας ε, με αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στον κανονισμό ελέγχου απλά και μόνο ευθυγράμμιση, προσαρμογή του, συστήμα, του κανονισμού ελέγχου στην επιτροπολογία και τους κανονισμούς και διατάξεις επιτροπολογίας μέσω της συνθήκης Λισαβόνας. Θα, θυμόσαστε ότι είναι ένας κανονισμός, κανονισμός που πρόσφατα εγκρίθηκε πολύ λίγο πριν σε σχέση με την έγκριση α, ε, της και πρέπει να υπάρξει αυτή η προσαρμογή. Θα θυμόσαστε ότι ο κανονισμός εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό ελέγχου που εγκρίθηκε το 2011, ο 404 του 2011 κανονισμός εγκρίθηκε προτού γίνει αυτό λόγω του ότι υπήρχε κατεπήγον όπως είχε συστηθεί τότε με σαφή τρόπο από την από τους ελεγκτές του ελεγκτικού συνεδρίου. Λοιπόν, Τούτου λεχθέντο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την πρόταση που είναι περίπλοκη ακολούθησε τι κατευθυντήριε γραμμέ που υιοθετήθηκαν, εγκρίθηκαν από τα θεσμικά όργανα για την προσαρμογή, για την τροπολογία όσον αφορά τα θέματα της συνθήκης Λισαβόνα. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι προσαρμόζουμε τα θέματα επιτροπολογία. Δεν προσθέτουμε κανένα νέο στοιχείο επί τη ουσία στον κανονισμό ελέγχου. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες αλλαγές καλύτερης διατύπωσης όσον αφορά τη νομική διατύπωση θεμάτων ή ανανέωσης διατυπωτικά της γλώσσας. Έχουμε εδώ την ε, κοινότητα που αντικαθίσταται από την Ένωση, ανάγκη που ήταν ε, επιτακτική να γίνει και έχουμε προσαρμόσει κάπως τον, την γλώσσα της διατύπωσης του κανονισμού με την αντίστοιχη ε, ορολογία που χρησιμοποιείται στις προτάσεις μας για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Το καλύτερο παράδειγμα είναι για αυτή την ανανέωση ορολογίας αντί μέτρα κατεπήγοντα κάνουμε λόγο για προσωρινά μέτρα προσαρμόζουμε με αυτόν τον τρόπο την ορολογία ώστε να προσαρμοστούμε με τις προτάσεις κανονισμού. Αυτά είναι τα δύο μόνα στοιχεία που εμπεριέχει αυτή η πρόταση. Προσαρμογή της διαδικασίας επιτροπολογίας και κάποιες αλλαγές, περιορισμένες αλλαγές για βελτιώσεις ή προσαρμογές γλωσσικές. Αλλά όχι αλλαγή επί της ουσίας. Όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης ή τις κατεντολήν πράξης ε, είναι περίπλοκος ο κανονισμός μια και υπάρχουν 34 άρθρα στα οποία μετατρέπουμε τις ε, διατάξεις ε, του κανονισμού ελέγχου σε πράξεις ε, εκτέλεσης, εκτελεστικές πράξεις. Υπάρχουν 11 άρθρα όπου την επιτροπολογία του σημερινού κανονισμού την μετατρέπουμε σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Και έχουμε και ένα τμήμα με μείγμα των δύο. Έπρεπε, ας το πω έτσι, να τα κεντήσουμε και να τα πλέξουμε με αυτόν τον τρόπο ώστε να συνδέουμε αυτές τις διατάξεις που αφορούν το ε, δικαίωμα, το δίκαιο που προσαρμόζεται και προβλέπει και πρόσθετες ε, διατάξεις όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και από την άλλη πλευρά για τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν ε, την αποσαφήνιση για να υπάρξει καλύτερος εναρμονισμός μεταξύ των κανόνων και διατάξεων που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Και εδώ περνάμε στις κατεξουσιοδότηση κατεντολή πράξη. Όπως βλέπετε σε σχέση με κάποια άρθρα αυτό που κάναμε είναι διαχωρίσαμε τις κατεξουσιοδότηση πράξη από τις ε, κατεντολήν πράξεις. Διότι υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις που παρουσιάζονται και μάλιστα και μέσα στο πλαίσιο ενός ιδίου τύπου ή μιας τυπολογίας. Πρόκειται για ένα περίπλοκο κανονισμό. Στο τέλος τέλος πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν 63 προτάσεις για κατεξουσιοδότηση πράξη και 22, ε, κατεντολήν πράξης και 22 ε, κατεξουσιοδότηση. Είναι σημαντικό εδώ η εξή ε, αποσαφήνιση. Όταν κάνουμε λόγο για εκτελεστικές πράξεις, ο σημερινός κανονισμός προβλέπει και έτσι αντανακλάται στη νέα πρόταση Κάποια, κάποιες 20 τέτοιες περιπτώσεις έχουμε όπου δεν συμπεριλαμβάνεται καμιά μορφή επιτροπολογίας. Αυτό δεν είναι καινούριο. Έτσι έχει στον υφιστάμενο κανονισμό. Και έτσι λοιπόν, θεωρώντας ότι όταν θα είναι αναγκαίο και είναι εφικτό, θα μπορούμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη διατήρηση της εντολής της Επιτροπής, που θεωρούμε ότι με βάση τον κανονισμό, τον ε, ουσιώδη κανονισμό, προβλεπόταν με βάση την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την καθημερινή ανάγκη να προσαρμόζουμε τεχνικές ε, διατάξεις ε, σε μια διαρκώς ε, ενρευστό ευρισκόμενη διαδικασία ελέγχου των αλλιευτικών δραστηριοτήτων της αλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία ζητούν μικρές τέτοιες αλλαγές ή προσαρμογές και θεωρούμε ότι ο κανονισμός ελέγχου πρέπει να έχει την αναγκαία αυτή ελαστικότητα ώστε μέσω κανονισμών δράσης άμεσης και τεχνικού χαρακτήρα να μπορεί να προσαρμόζεται όταν ζητείται αυτό από τα κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι πραγματικά όσον αφορά την ε, περίπτωση κατεκτέλεση πράξεων εφαρμόζουμε τα όσα προβλέπονται από το 182 κανονισμό του 2011 στο άρθρο 5 την τακτική δηλαδή διαδικασία και την κατεξουσιοδότηση της κατεξουσιοδότηση πράξης έχουμε εντολή χωρίς ε, περιορισμό χρονικό. Αυτή είναι απλά η πρόταση που υποβάλαμε. Όπως γνωρίζετε όμως καλύτερα από μένα εσείς σε αυτό το θέμα για τις κατεξουσιοδότηση πράξης ή για την εντολή της Επιτροπής να συντάσει τέτοιες ε, πράξεις αν αυτό είναι περιορισμένο ή όχι στη διάρκεια του χρονικά όπως και σε άλλες περιπτώσεις προχωρήσαμε στη συζήτηση σε σχέση με τα θέματα της συνθήκης της Λισαβόνα και προτείνονται λύσεις όπως για παράδειγμα τριετής διάρκεια ή ανανεώσιμη εντολή και έτσι λοιπόν επ' αυτού πρέπει να διαφοροποιήσουμε και να πούμε ότι μια και έχει δείξει το μέτρο της ελαστικότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας αυτών των εντολών θα πρέπει η ίδια ελαστικότητα να μπορεί να ισχύσει μέσα στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού τελικά. Και εν κατακλείδη αυτό που προτείνει προτείνουμε με αυτές τις αλλαγές είναι να δοθεί μια νομική κάλυψη για τις διατάξεις που έχουμε στο σημερινό κανονισμό και την εφαρμογή του στο 404-2011 πρόκειται για κάποια μικρή τροποποίηση όμως της νομικής βάσης σε σχέση με αυτά που γίνονται με τον κανονισμό 404. Δεν χρειάζεται σε αυτόν τον κανονισμό να αλλάξει όμως ε, από το αναγκαίο ή σε βάθος ο κανονισμός αυτός 404-2011. Πρόκειται λοιπόν για μια λησβονοποίηση, προσαρμογή σε σχέση με την ε, συνθήκη Λισαβόνας όλων αυτών των λεπτομεριών. Δεν έχουμε κάποιο νέο στοιχείο ενώπιόν μας ε, σε σχέση με το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης. Ίσως είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση φάση αυτή τη στιγμή. Προσαρμόζουμε στι συνθήκε τη αγώνα κάποια πράγματα. Αν υπάρχει κάποια δικαιολογία για την αλλαγή σε βάθο ε, διατάξεων ελέγχου μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, αυτό θα απορρεύσει από το θέμα τη ε, μεταρρύθμισης τη ίδια. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε και να δούμε αν κάποιες αλλαγέ είναι πράγματι αναγκαίε σε ευρύτερο, σε ευρύτερο πλαίσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια κυρία Τόμα έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στους στόχους αυτής της προσαρμογής της συνθήκη της, της Γενικά αυτή η ευθυγράμμιση έχει ως στόχο τη βελτίωση της ε, διακυβέρνησης και άρα και του τρόπου εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής αλλίας. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει βελτίωση, εναρμόνιση ε, ε, στον τομέα των ελέγχων. Και προκειμένου η έλεγχη να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι δίκαιη και ισότιμη. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και πιο αποτελεσματικοί. Τώρα, συγκεκριμένα, θα λάβουμε θέση στα εξή ζητήματα. Προτείνεται περίπου 60 μέτρα, πολύ διαφορετικά, από τη ζήγηση μέχρι το μορφότυπο, μέχρι και την απαγόρευση αλίας σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή πολλά πολλά και διαφορετικά μέτρα. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε έναν τρόπο λήψης αποφάσεων και θα δούμε ποια θέση θα λάβει η Επιτροπή. Με ποιον τρόπο λοιπόν επιλέγουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο απόφασης. Στα άρθρα 17 και 21 προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισμένα είδη σκαφών σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ε, γιατί εδώ να ζητάμε σε πράξη και όχι άλλη μέθοδο. Έγιναν διαβουλεύσεις καροετοιμασίας σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, λέτε. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Πότε έγιναν, ποιοι συμμετείχαν, ποια ήταν η διάρκεια τους και κυρίως εάν τα ΡΑΚ θα συμμετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Δεύτερο σημείο. Λέτε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην ουσία του βασικού νομοθετικού κειμένου. Αλλά, εάν συγκρίνουμε το αρχικό κείμενο Πράγματι δεν υπάρχουν αλλαγές στην ουσία, αλλά το νέο κείμενο πηγαίνει σε ένα βαθμό λεπτομέρειας που δεν τον είχε ο αρχικός κανονισμός. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένας τρόπος να υπάρξει μεγαλύτερη ομοιογένεια Όσο περισσότερο εξετάζουμε τις λεπτομέρειες και ρυθμίζουμε τις λεπτομέρειες, τόσο μεγαλύτερη εναρμόνιση πετυχαίνουμε. Ένα παράδειγμα για αυτό που μόλις είπα. Άρθρο 92 με βάση το οποίο ρυθμίζεται η απόδοση μορίων ποινή σε περίπτωση παραβίασης. Εδώ λέγεται λοιπόν ότι για την ίδια παράβαση θα πρέπει να αποδίδονται τα ίδια μόρια. Ίσως καλύτερα να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και να ρυθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλονται αυτά τα μόρια ποινής. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ κυρία Τόμας. Ε, κυρία Φράγα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα μια σειρά ερωτήσεων να διατυπώσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με θέματα αυτού του κανονισμού και κάποια σχόλια να κάνω. Πρώτα απ' όλα για την προσαρμογή που γίνεται σε σχέση με το αντί να λέμε κοινότητα, ένωση κτλ. Δεν είναι μόνο σε σχέση με τα άρθρα για το 2 ή και άλλα, δεν εμπεριέχεται εκεί. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα τα σημεία με τον ίδιο τρόπο ενιαία αυτή η προσαρμογή. Δεύτερο, σε σχέση με το άρθρο 7 στο εδάφιο 5 Υπάρχει ένα έξι που θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εδώ γίνεται ειδική αναφορά σε σχέση με τα θέματα των μικρών σκαφών των αλλιευμάτων όταν στο αρχικό κείμενο δεν γίνεται αυτή η διαφοροποίηση εγκρίσεις εκφόρτωσης δηλαδή σε σχέση με μικρά σκάφη. Στο άρθρο 9, στο σημείο 10, εδάφιο 10, στο σημείο α, υποχρέωση να υπάρχει δυνατότητα εξοπλισμού, δορυφορικού εντοπισμού ε, των σκαφών. Με αυτό τι σημαίνει, ότι μέσω του, των κατεξουσιοδότης συμπράξεων θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ε, για τα κάτω από ε, μέχρι 12 μέτρα σκάφη και για το επόμενο ε, δεν συμφωνώ με την ε, διαφοροποίηση της διαφοροποίησης με τις κατεντολήν πράξεις και κατεξουσιοδότηση πράξης. Θα είναι κάτι το οποίο όμως πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι κατεκτέλεση πράξης πρέπει να είναι το μεγαλύτερο μέρος. Στο 55 εδάφιο 4 θα ήθελα να μου πείτε γιατί η συγκεκριμένη διαβούλευση σε σχέση με την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή έχει διαγραφεί. Γιατί έχει διαγραφεί αυτό το στοιχείο και δεν συμπεριλαμβάνεται πια. Και επίση θα ήθελα να μου πείτε γιατί στο άρθρο 58 στο 7ο εδάφιο έχουν τα όσα προβλέπονται για την ιχνηλασιμότητα και τους ελέγχους ιχνηλασιμότητας αλλιευμάτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Θέλω να ξέρω τι συνέβη σε σχέση με τα θέματα αυτά ιχνηλασιμότητας. Αυτά νομίζω ήταν και στη συνέχεια μια στιγμή έχω και διαφορετικές απόψεις για κάποια άρθρα για το 1-2 π.χ. όπως είπε η κυρία Τομάς εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι θέμα εκτέλεσης και όχι κατεξουσιοδότηση πράξης. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί διότι είναι σημαντικό. Ο εναρμονισμός είναι νομίζω κάτι που πρέπει καλύτερα με τις κατεξουσιοδότηση πράξης να καλύπτεται. Και για την προθεσμία ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται ε, κάποια αλλιεύματα με ασφάλεια προσαρμόζεται η ασφάλεια, η προθεσμία σε 15 ημερών. Τι γίνεται εδώ με την κατεντολή ε, ε, πράξη. Αυτά ήταν τα όσα είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω από πλευράς μου ότι μόνο σε κάποια θέματα θα ήθελα να περιοριστώ από αυτή την έκθεση αυτή η έκθεση αφορά η Υποτίθεται ότι αφορά μικρές προσαρμογές ε, διατυπωτικές και όχι μεγαλύτερες. Γι' αυτό θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε αυτές τις πτυχές, ε, να πω ότι αυτός ο, αυτή η πρόταση κανονισμού αφορά επίσης ε, και κάποιες ε, διατάξεις που εδώ και χρόνια τώρα όταν αρχίσαμε να ε, έχουμε επαφές ε, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ελέγχου στο ΒΙΓΟ, ρώτησα αν υπήρξε πολιτική πίεση που ασκήθηκε για να μπορέσουν κάποια πράγματα να εγκριθούν. Δηλαδή πίεση, ας το πω έτσι, σε σχέση με τους δημοκρατικούς ε, κανόνες και διατάξεις ε, όσον αφορά τον έλεγχο, αν αυτό περιόριζε ή όχι το έργο και αν αυτά αντανακλώνται σε κάποιες αρχές ε, και μετά από πέντε ή έξι χρόνια μιας κοινή αλλιευτικής πολιτικής όταν τοποθετήθηκε διευθυντής για τους τα καθήκοντα ελέγχου και ο έλεγχος από Επιτροπής της Βαλτικής. Ένα παράδειγμα πρέπει να δώσω από τη δική μου τη χώρα, την Πολωνία, για να γίνει κατανοητό. 11.000 φορές ασκήθηκαν τέτοιοι έλεγχοι σε σχέση με εμά. Εντάξει, στην Φινλανδία 50 όλοι και όλοι οι έλεγχοι. Πώς γίνεται αυτό. Και να στα επαναλάβω άλλη μια φορά για να, γίνει, να γίνουν πιο κατανοητά. Εμείς 11.000 φορές ελεγχθήκαμε ως Πολωνία. Η Φινλανδία 50 φορές όλες και όλες. Ας το σκεφτεί κανείς αυτό και ας προβληματιστεί να δει γιατί υπάρχει τέτοια τρομακτική δυσαναλογία στους όρους. Η επεξήγηση δεν είναι σίγουρα εύκολη. Δεν υπάρχει εύκολο επιχείρημα για να δικαιολογήσει κανείς κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό αρνητική διακριτική μεταχείριση κάποιων εμπλεκόμενων. Δεν είναι κάποιος περιορισμός ε, του ανταγωνισμού, στρέβλωση του ανταγωνισμού αυτή η κατάσταση ή όχι. Συνέβη αυτό έτσι, είναι γεγονός. Τα στοιχεία, τα δεδομένα το λένε αυτό. Είναι αδιαμφισβήτητα. Τι γίνεται λοιπόν με τους ελέγχους. Πραγματικά πρόκειται δηλαδή για θεμητό πλαίσιο ελέγχων με τέτοιες διαφορές. Πρόκειται για σεβασμό των νομικών και ε, ρυθμίσεων και διατάξεων. Αλλά τέλος πάντων σε σχέση με άλλες χώρες ας μην ε, τις στριμώξουμε με τέτοιο τρόπο. 11.000 παράδειγμα Πολωνία, 50 έλεγχοι Φινλανδία. Ε, είναι μια πολύ ακραία κατάσταση που διαμορφώνεται όσον αφορά τους ελέγχους. Αυτό το σύστημα, αν με αυτόν τον τρόπο συνεχιστεί και έτσι χαρακτηρίζεται με τέτοια στοιχεία και στρέφομαι προς τον κύριο Διευθυντή, και πρέπει να ζητήσουμε να ασκηθεί η επιρροή του ώστε στο μέλλον να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μην καταλήγουμε σε μια τέτοια κατάσταση εκ νέου. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό ώστε να μην έχουμε τέτοια αριθμητικά στοιχεία, τέτοια στρέβλωση, τέτοια αδικία που να έχουμε μια, ένα τόσο δυσανάλογο τρόπο ελέγχου. Σας ευχαριστώ κύριος Πένας της Επιτροπής μπορεί να σας δώσει απάντηση για αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρέπει να πω για τις παρεμβάσεις που καταδεικνύουν ότι πραγματικά με όλες τις προσπάθειες που κάναμε υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κατηγοριοποίηση κάποιων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ή κατ' εντολή είναι συζητήσιμα θέματα. Είναι σαφής η κατ εντολη ειναι συζητησιμα θεματα ειναι σαφη η φιλοσοφια που μας εμπνέει. Πάντα όταν υπάρχουν πράξει, πρέπει διατάξεις ή πρόσθετες ε, ε, τέτοιες ε, πράξεις πρέπει να είναι κατ' εξουσιοδότηση πράξης και πρέπει όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο να εκτελούν αυτές τις πράξει, χωρίς να υπάρχουν όταν δεν υπάρχουν νέε υποχρεώσει, είναι κατ' εκτέλεση πράξει. Είναι σαφή η θεωρία και στην πρακτική εφαρμογή λογικό να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις θεών ζωνών που δεν είναι σαφείς και πρέπει αυτό να θεωρηθεί ένα θέμα που μπορεί να τεθεί σε συζήτηση. Δεν θέλω να επισέθω σε λεπτομέρειες, αλλά η Επιτροπή δεν έχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτή την, αυτές τις προσαρμογές και τη ρύθμισή τους. Η κατεξουσιοδότηση πράξης ε, είναι, έχουν μια συνιστόσα, στο πω έτσι, διοικητική που είναι πιο επιβαρημένη, επιβαρύνεται περισσότερο. Και αν εσείς οι συνομοθέτες του Συμβουλίου ως Ευρωκοινοβούλιο θεωρείτε ότι είναι προτιμητέο να είναι κατεκτέλεση πράξης, ε, τότε δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα να ε, διαλύσει την κατάσταση πραγμάτων. Τώρα, για το αν υπήρξε διαβούλευση των ε, επαϊόντων ή των ράξ, δεν υπήρξε τέτοια διαβούλευση. Για ένα απλό λόγο, γιατί αυτό είναι ένα θέμα νομικού χαρακτήρα, όπου θεωρούμε ότι οι οργανισμοί διαβούλευσης που έχουμε και λειτουργούν, θεωρούμε ίσως ότι δεν ήταν απαραίτητο να διαβουλευτούν αυτοί επ' αυτού του θέματος που δεν είναι ουσιώδες και είναι κυρίως έχουν χαρακτήρα διοικητικό ή διοικητικών προσαρμογών και θεωρήσαμε ότι η ομάδα επαϊόντων και τα ράξα δεν ήταν το πιο εύθετο θέμα να ασχοληθούν με αυτό. Έχουν ήδη υπερβολική δουλειά και ασχολούνται με άλλα θέματα. Αληθεύει λοιπόν ότι δεν διαβουλευτήκαμε με αυτούς για αυτό το θέμα. Τώρα πάλι σε σχέση με τις ερωτήσεις της κυρίας Φράγκα. Πράγματι πιστεύω ότι ε, όσο αφορά την ε, ε, εξαίρεση μήκους διαστάσεων ε, σκάφους ε, είναι κάτι που καταρχήν δεν μπορεί αυτό να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να είναι κατεξουσιοδότηση πράξη και μπορεί να συζητηθεί αυτό. Όμως η βασική μας φιλοσοφία είναι σαφής για το πώς πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Για το SPCF είναι, ανταποκρίνεται σε μια θέση που, τοποθέτηση που υιοθετήσαμε μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και αναφέρεται στο γεγονός ότι οι νομομαθείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμένουν και επιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαφυλάξει το δικαίωμα ανάληψη ιδία πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτική διαβούλευση με κανέναν προτού εγκριθούν κάποιε προτάσει ή αναλυφθεί πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι υπήρξε η προσπάθεια να αποφευθεί αυτή η πτυχή πριν από την οποιαδήποτε δηλαδή έγκριση πράξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προβλέπεται υποχρεωτική διαβούλευση με κανέναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο αυτό της ε, ε, κοινή αλληλευτικής πολιτική ή των προτάσεών μας. Για ε, την προθεσμία 15 ημερών μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ τελεσίδικα τώρα. Το μόνο θέμα που ε, τίθεται είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει δεν θα χρειαστεί αυτόνομα να γίνει σε σχέση με τον κανονισμό. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, να εξετάσουμε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και σε συνάρτηση με αυτό το σημειώνω για να σας απαντήσουμε. Προτιμώ να μην απαντήσω αυτοσχεδιάζοντας τώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν θα μπορεί ή θα πρέπει να τροποποιείται η προθεσμία 15 ημερών. Σε σχέση με την παρατήρηση του κυρίου Κροβάρσικ, ε, εννοώ ότι δεν ε, συνδέεται άμεσα με αυτή την πρόταση κανονισμού, όμως θα ήθελα να δώσω απάντηση, Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ανέφερε και είναι αυτά τα θέματα πολύ σπουδαία. Προσέξτε, εγώ μεταξύ άλλων πραγμάτων είμαι και εγώ συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της, του σώματος αυτού και μέσα σε αυτό το σώμα υιοθετούνται τα κοινά προγράμματα ελέγχου και για τη Βαλτική όπως γνωρίζετε και εκεί αναλύονται επακριβώς ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, ποιοι έλεγχοι και πόσοι θα γίνονται σε κάθε περιοχή ή ζώνη και όλα αυτά βασίζονται σε τεχνικού χαρακτήρα στοιχεία όπως και την αξιολόγηση κινδύνων π.χ. Υπάρχει έργο υποεκτέλεση και εξέλιξη για την αξιολόγηση κινδύνων. Γίνεται εκεί, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι εκεί όπου υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μηχανισμών που διασφαλίζουν ότι οι προτεραιότητες για τους ελέγχους έτσι θα θεσπίζονται και θα ιεραρχούνται και για την ε, ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων, αλλά όχι αυθαίρετα. Μπορώ να διασφαλίσω τον κύριο ότι σε όλες τις συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής του ε, Οργανισμού Ελέγχου ε, στο Βίγο, όλα αυτά τα οποία εκεί συζητώνται, μπορώ να σας διασφαλίσω ότι ποτέ δεν υπήρξε παράπονο από πλευράς κάποιου κράτους μέλους. Ότι δηλαδή τα σχέδια ελέγχου το, του οργάνου ελέγχου στο Βίγο ήταν αυθαίρετα ήταν αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Πάντα λειτουργούν υπό το πρίσμα της αξιολόγησης κινδύνων και ποτέ αυθαίρετα ή ασίδωτα. Και μπορώ να σας διασφαλίσω ότι ούτε ο Πολωνός αντιπρόσωπος ποτέ παραπονέθηκε όπως δεν παραπονέθηκε και κανείς άλλος από άλλο κράτος. Σας ευχαριστώ κυρία Φράγκα παρακαλώ. Για το 58 σε σχέση με την ανιχνευσιμότητα. Μπορεί να διευκρινίσει η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ εγώ. Αυτές οι δύο διατάξεις, το 58, 7α και 7δ, προσθέθηκαν ώστε να έχουμε μια απόλυτα σαφή νομική βάση για αυτές τις ε, ε, διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις βρίσκονται στον εκτελεστικό κανονισμό 404-2011. Ε, Εκτελεστικές διατάξεις δεν είναι τίποτα το καινούριο το οποίο εισάγεται. Αυτά τα αναφέρω για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί, αυτές οι εξαιρέσεις είναι θεμητές. Αυτές έχουν μεταφερθεί και ενταθεί στην λησβονοποίηση του κανονισμού. Τέσσερις οι ίδιες διατάξεις με επιθυμία των ίδιων των κρατών μελών εντάχθηκαν σε αυτό το σημείο με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Euh, euh, δεν ξέρω αν θα το κλείσουμε τώρα το θέμα, αλλά γιατί από ό,τι φαίνεται παραμένουν πολλά ακόμα ανοιχτά ζητήματα. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Πένια μας εξήγησε πώς επιλέγεται μεταξύ κατεξουσιοδότησης και εκτελεστικών πράξεων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπήρχαν ε, κριτήρια νομικής φύσεως, για παράδειγμα όταν αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, τότε θα έπρεπε ε, η δημόσια διοίκηση των κρατών αυτών που έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητε να συμμετέχει στη λήψη τη απόφαση. έτσι δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο που έχει ζητήσει το λόγο. Ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα, στο 12, για την αντιπροσωπεία μας στην Ιρλανδία. Ξέρετε ότι ε, έγινε μια επίσκεψη από τις 12 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσα και εγώ να σας ενημερώσω, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλαχερ για να μας κάνει μια καλύτερη παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε στείλει μια πολύ πλήρη έκθεση της ε, αποστολής μας μπορώ να πω για τους συναδέλφους που είναι εδώ και κυρίως εκείνους που δεν είναι εδώ, ότι όταν ε, λάβαμε την απόφαση για την ε, συμμετοχή στην αποστολή, είδαμε ότι όλοι θέλουν να πάνε. Καθώς πλησιάζει λοιπόν η ημερομηνία της αποστολής, ε, τα μέλη ίσως για πολύ, πολύ ορθούς λόγους αρχίζουν να λένε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν και αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί την τελευταία στιγμή έχουμε ακυρώσεις. Βέβαια, αναγνωρίζω ότι ε, ο λόγος μπορεί να ήταν ανωτεραβία, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν τελικά στην ε, αντιπροσωπεία και θέλω να, ε, τους κύριους Ρόντες και Στέβενσον και θέλω να σας ευχαριστήσω και σας κύριε Πρόεδρε για την υποστήριξη. Εν πάση περιπτώσει, η τριμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας επισκέφθηκε την Ιρλανδία και ίσως να ήμασταν τρεις, αλλά ούκον το πόλο το F. Συναντήσαμε αντιπροσωπείες ε, αλλιέων από τον τομέα της πελαγικής ε, αλίας και επισκεφτήκαμε το Χίλιμπεκ, μάλλον, μια σημαντική περιοχή για την ε, αλληλία, από την οποία κατάγομαι κιόλα. Συναντήσαμε εκπροσώπους των ψαράδων από την περιοχή αυτή, τους ε, ικανοποίησε ιδιαίτερα το γεγονό ότι τους ε, συναντήσαμε και μιας και είχαμε συζητήσει και το θέμα τον Απρίλιο, στο, στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν, δεν υπάρχει πρόεδρος. Αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία υιοθέτησαν την νομοθεσία για τις κυρώσεις. Η κυρία Θαμανάκη γνωρίζει την θέση μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί στο ρόλο που θα πρέπει να έχει αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Όταν συζητάμε για την αναθεώρηση της πολιτικής αλίας, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την βιομηχανία αλίας ε, ότι στο μέλλον θα φροντίσουμε τα συμφέροντά μας αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε καν το παρόν και δεν έχουμε την νομοθεσία την κατάλληλη στη διάθεσή μας. Εν πάση περιπτώσει, συνολικά ήταν αρκετά χρήσιμη η συνάντηση στο Κίλιμπεξ και γενικά στην Ιρλανδία. Συναντήσαμε παραγωγούς αλληλείς επισκεφτήκαμε ένα εργοστάσιο ε, μεταποίησης σκουμπριού και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ποιότητα από τη στιγμή που εκφορτώνεται το αλίευμα από το πλοίο μέχρι το τέλος. Επίσης συναντηθήκαμε με ψαράδες από τις παράκτιες περιοχές. Εχθές που συζητούσαμε τις στράτες αναφέρθηκε πρέπει να μην αγνοήσουμε τους μικρούς βιοτέχνες αλληλείς. Επίσης ε, επισκεφτήκαμε ένα πλοίο στην Προβλήτα μενθοπελαγικής αλίας και είδαμε από κοντά τα προβλήματα που έχουν όταν αλλιεύματα από ευρωπαϊκά πλοία αλλιεύονται στον Ατλαντικό. Για παράδειγμα, σκουμπρία αλλιεύεται στο Ατλαντικό, πολύ διαφορετικά μεγέθη και πολύ πολύτε. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία έχουν έναν τρόπο να επιλέγουν ρίχνοντας το βυθό πίσω τα άλλα ψάρια και τελικά καταλήγουν να ψαρεύουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Αυτό είναι καταστροφικό για τον πληθυσμό. Πρέπει να αναλάβουμε δράση εδώ και η Επιτροπή ιδιαίτερα. Εάν ένα σκουμπρί συγκεκριμένου μεγέθους έχει υψηλότερη τιμή, και επιλέγεται αυτό και τελικά πετιούνται στη θάλασσα πίσω, εδώ έχουμε πρόβλημα. Θα έπρεπε ανταυτού να εκφορτώνονται τα αλλιεύματα που όντως αλλιεύτηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία στην Ιρλανδία. Κύριε Στέβενσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατ Δεκόουπ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη και στο Κίλιμπεγκς και στην ευρύτερη ζώνη του Γκόλουεϊ. Σας πω μια μικρή ιστορία εδώ. Όταν συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους των μικρών αλλιέων από τα νησιά από το Άραν Μόρ, Ίνις Μόρ κτλ. Η αντιπροσωπεία των Αλλιέων είχε σαν ηγέτη έναν ιερέα. Και μάλιστα είχε πάρει ένα τηλέφωνο το οποίο του έλεγε ότι ο Πατ The Κόουπ είχε παρετηθεί αλλά βέβαια μπερδεύτηκε διότι δεν είχε παρετηθεί ο Κόπ αλλά ο Pope, ο Πάπας. Και έτσι ησύχασε ο ιερέας από τις νήσους Άραν. Η κατάσταση επίσης και σε σχέση με τις πελασγικές αλλιευτικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Ένα από τα στοιχεία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι το 88% των αλλιευμάτων ε, στα Ιρλανδικά ύδατα δεν τα συλλέγουν Ιρλανδοί αλλιείς. Οι ανοιχτέ θάλασσε, λοιπόν αλλιευτικέ δραστηριότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές, τις έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ μεγάλα Ολλανδικά σκάφη που έχουν τις ίδιες ποσοστώσεις με τους Ιρλανδούς. Οι Ιρλανδοί ολοκληρώνουν την αλία σκόμβρου σε τέσσερις μήνες, ενώ οι Ολλανδοί με την ίδια ποσόστοση το κάνουν σε δώδεκα μήνες. Είναι περίεργο, Επιξεργάζονται βέβαια τα λιεύματά τους εντός του σκάφους, έχουν ε, δυνατότητες μέτρησης ε, των ε, ταξινόμησης των αλλιευμάτων εντός και ταυτόχρονα βέβαια απορρίπτουν 9.000 τόνους σε αιτήσια βάση. Αυτό είναι απαράδεκτο και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2014 μετά από την ψηφοφορία μας θα απαγορευτεί στα πελασγικά ήδη η απόρριψη πλήρως. Και επίσης και η εγκατάσταση ε, κάμερας ε, θα ε, δίνει την δυνατότητα να βελτιωθεί η κατάσταση, να ελέγχεται καλύτερα. Πάντως παναλαμβάνω ότι το θέμα των ίσων Φερόε και της Ισλανδίας δεν έχει επιληθεί ακόμα Υποτίθεται ότι εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, ακολουθήσαμε την κατεπίγουσα διαδικασία. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος που συναντηθήκαμε στο Κίλιμπεξ αναρωτιέται «Μα τι κάνετε, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα μέσα τα οποία ε, έχετε, δεν χρησιμοποιούνται τα μέσα τα οποία έχει η Επιτροπή, έχετε δώσει στην Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί η εγκληματική εμπάση περιπτώσει δραστηριότητα των αλλιέων από την Ισλανδία και τα νήσους Φερόες. Είναι λοιπόν σημαντική η επίσκεψη αυτή και το Ινστιτούτο της Θάλασσας στο Galway είναι από τα πιο σημαντικά και άξιζε την επίσκεψη εγώ έκανα μια ομιλία σε ένα αντίστοιχο τέτοιο Ινστιτούτο στο Άμπερσουετ στη Σκοτία και μπόρεσα να συγκρίνω το τι κάνουν τα δύο Ινστιτούτα και καλό θα ήταν να υπήρχε μια πιο επίσημη σύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητες τους. Ίσως να τα συζητήσω ε, σε έφθετο χρόνο αυτά με τον Πατ Δεκόουπ. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον, η κυρία Ρόντοστ. Ναι και στην τελευταία μας συνεδρίαση Ευχαρίστησα τον κύριο αυτό και ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ χρήσιμη αποστολή και είναι πολύ όμορφη και η χώρα και όποιος δεν συμμετείχε σε αυτή την αποστολή έχασε πραγματικά. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία περιγράφηκαν δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο όμως με συγκλώνησε είναι ότι οι Ολλανδοί μόνο 300 γραμμάρια έχουν τα οποία ε, οδηγούν στην εκφόρτωση. Πράγμα αυτό που δείχνει ότι εδώ υπάρχουν εγκληματικές ε, πράξεις ε, και προηγούμενα αναφέρθηκαν τα σχετικά. Επίσης μας πληροφόρησαν ότι υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές στο πλοίο που είναι πολύ χρήσιμες αλλά δεν επαρκούν επίσης ε, μπορούν να χειραγωγήσουν και να πειράξουν αυτές τις μηχανές ώστε να μην λειτουργούν όπως πρέπει. Και εδώ θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί επικοδομητικά θετικά η παρακολούθηση με ε, κάμερες. Μας είπαν όμως ότι δεν είναι κανένα πρόβλημα να τις πειράξουν λέει. Και υπάρχει θερμή παράκληση κυρίως για τα μεγάλα ε, σκάφη, πρόσθετα παρατηρητές να βρίσκονται ε, στο ίδιο το σκάφος. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με αυτούς τους ελέγχους για αυτές τις δραστηριότητες. Πρέπει να προβληματιστούμε σε βάθος σοβαρά, να δούμε πώς θα διοργανώσουμε αυτούς τους ελέγχους. Ήταν πολύ σκανδαλώδη όλα αυτά, τεράστιο σκάνδαλο αυτά που μας είπαν επί τόπου. Και πραγματικά η ζημιά είναι τεράστια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρόντος επαναλαμβάνουμε το αίτημα και την τοποθέτηση προς τον κύριο Γκάλαχερ. Ευχαριστίες μας. Λίγη συνεδρία θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ. No, that is very cool, I think. That's awfully No, this, I was complaining